Ladies and gentlemen, please be seated. Κυρίες και κύριοι, καθίστε παρακαλώ. Um, good afternoon. Uh, I'm... Καλησπέρα σας. Χαίρομαι και είμαι και βεβαίω ότι χαίρεστε κι εσείς που βρίσκεστε εδώ. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν συζητήσεις σε καλό πνεύμα. Συγγνώμη για τη βραχνάδα στη φωνή μου, θυμίζω το Λουίς Άρμστρονγκ, αλλά θα προσπαθήσω να μιλάω λίγο πιο δυνατά. Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι η συνεδρίασή μας μεταδίδεται ζωντανά στο διαδίκτυο, ως συνήθως. υπάρχει διερμηνία κατά προτεραιότητα για τα μέλη της Επιτροπής ε, Ασφάλειας και Άμυνας και πριν σας ζητήσω να κρίνετε την ημερήσια διάταξη θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι πρέπει να διαγράψουμε το σημείο 3 αφού αλλάξουμε και τη σειρά των σημείων, Το πρώτο ουσιαστικό σημείο είναι η συζήτηση για την έκθεση του κυρίου Πάσκου εφαρμογή της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, ετήσια έκθεση. Κατόπιν έχουμε τα αποτελέσματα της διάσκεψης του ΝΑΤΟ και το τρίτο σημείο επρόκειτο να το παρουσιάσει ο κύριος Ούρμας Πάετ για την πρώτη συζήτηση για την έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση Άμυνας. Ε, όπως θα γνωρίζετε βέβαια περισσότεροι από εσά, ο κύριος Πάετ αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα υγείας Ευτυχώς βέβαια αναρώνει, αλλά πρέπει ακόμα να παραμείνει κλινίδης, επομένως αναβάλλεται το σημείο αυτό. Το χρονοδιάγραμμα όμως έγκρισης της έκθεσης θα παραμείνει, επομένως παραμένει η ίδια προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Η 7η Σεπτεμβρίου ήταν η ημερομηνία. Έχουμε λοιπόν δύο σημεία προσυζήτηση στην ημερήσια διάταξη. Η ετήσια έκθεση βάση της έκθεσης του Συμβουλίου για την εφαρμογή της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Η συγητής είναι ο κύριος Ιωάνν Μίρτσια Πάσκου και στη συνέχεια τα αποτελέσματα και οι κύριες αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Βασοβία θα μας τα παρουσιάσει ο αναπληρωτής ε, Γενικός Διευθυντή για Πολιτικές Υποθέσεις και ο κύριος Κώστερ, ο οποίος είναι γνωστός σε εσάς σας, ε, και ο πρόεδρος ε, του CMPD, του Τμήματος Διαχείρισης Κρίσεων και Σχεδιασμού, ο κύριος Γκάμπορη Κλόντι. Εάν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, εγκρίνεται η μερίσια διάταξη και χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση προτείνω να ξεκινήσουμε τις ε, παρουσιάσεις Έχουμε το πρώτο σχέδιο έκθεσης για την εφαρμογή της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας από τον κύριο Πάσκου. Οι πολιτικές ομάδες έχουν ορίσει και οδησίγητες, επομένως ε, μπορούμε να ε, συζητήσουμε την έκθεση αυτή. Κύριε Πάσκου, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε και τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε πρώτα το δικό μου το θέμα στη συνεδρίαση, γιατί και εγώ έχω κάποια άλλη υποχρέωση ε, και ήθελα να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα, το οποίο ούτως ή άλλως ήδη μας πιέζει. Όπως ε, γνωρίζετε, η έκθεση αυτή και η έκθεση του κυρίου Μπροκ επρόκειται να παρουσιαστούν νωρίτερα, αλλά δεδομένων ε, των συνθήκων ε, που δεν μπορούσαμε να τις αποφύγουμε, χρειάστηκε να αναβληθούν. Αυτό σημαίνει ότι οι εκθέσεις βρίσκονται εκ παραλλήλου με τα όσα συμβαίνουν ε, στο θέμα αυτό. Και όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, αλλά και όσον αφορά την πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Η έκθεση αυτή βασίζεται στην προϋπόθεση ότι λόγω των πρόσφατων εξελίξεων και το γεγονός ότι συσσωρεύονται οι προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, χρειάζεται διεξοδική αναθεώρηση της κοινής μας συναντήληψης ε, περί του τίνος πρόκειται όταν συζητάμε κοινή πολιτική ασφαλείας και άμυνας. Και έχουμε κυρίω θέματα διαχείρισης ε, κρίσεων και κυρίω κρίσεων εκτό Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αν θυμάστε, κυρίω στην ουσία τη έκθεση ασχολούμαστε με τι διάφορες επιχειρήσεις. Αυτή τη φορά θεωρήσαμε ότι δεδομένου ότι ασφάλεια είναι τόσο σημαντικά και στα μάτια των Ευρωπαίων πολιτών, δεδομένων και των τελευταίων αρνητικών ε, γεγονότων, ε, τρομοκρατία, μετανάστευση και ούτω καθεξής. Φαντάζομαι ότι γνωρίζετε ότι πρέπει να συμπληρώσουμε λίγο την αντίληψη που είχαμε, τα οποία ήταν κυρίως θέματα διαχείρισης κρίσεων, με θέματα ασφάλειας και άμυνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς μπορούμε λοιπόν να προσδώσουμε ουσία στο θέμα αυτό. Αυτό είναι κάτι το οποίο Όπως αντιληφθήκαμε άλλωστε και χθες στην Πρατισάβλα, ε, Σλάβα, το έχει αποδεχτεί, είπατε, εκπρόσωπος ε, και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, συντάσσονται έγγραφα, συζητώνται, εγκρίνονται για το θέμα αυτό. Γι' αυτό άλλωστε και έλεγα ότι η έκθεση ε, γίνεται εκ με τα όσα συμβαίνουν στον τομέα. Ξεκίνησα λοιπόν λέγοντας ότι η Ευρώπη δεν ελέγχει πλέον το περιβάλλον ασφαλείας της. βρισκόμαστε αντιμέτωποι με κρίσεις οι οποίες πολλαπλασιάζονται και γίνονται και πιο περίπλοκες. Και δεν έχουμε πλέον την πολυτέλεια να αποφασίσουμε πότε και πώς θα δράσουμε. Πρέπει να απαντάμε όσο καλύτερα μπορούμε σε αυτές τις προκλήσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της στρατηγικής της κυρίας ε, Μογκερίνη ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζουμε έναν ολόκληρο κύκλο κρίσης που σημαίνει ότι πρέπει να δούμε θέματα πρόληψης, εξέλιξης και σταθεροποίησης και επίσης τη δέσμευση ε, να αποφύγουμε, ε, να αποδεσμευτούμε από όλα αυτά πρόημα που είναι αυτό το οποίο ήταν πάγια πρακτική μέχρι τούδε βάσει της έκθεσης η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας θα πρέπει να βασίζεται σε μια βασική αρχή άμυνας, ε, αποτελεσματική χρηματοδότηση και πλήρη συνεργασία με τον ΝΑΤΟ. Υποστηρίζουμε λοιπόν την ανάπτυξη μιας τομεακής στρατηγικής ε, σε συνέχεια της στρατηγικής που παρουσίασε η κυρία Μογκερίνη και η κυρία Μογκερίνη μάλιστα επιβεβαίωσε και χθε στην Πρατισλάβα ότι Υπάρχει ήδη συγκεκριμένο επίπεδο φιλοδοξίας, συγκεκριμένα καθήκοντα, απαιτήσει και ε, προτεραιότητες για δυνατότητες οι οποίες ε, πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να επιτευχθεί αυτή η φιλοδοξία. Επικροτώ και το σύμφωνο ασφαλείας που πρότεινε η Γερμανία και η Γαλλία, διότι πολλές από τις ιδέες ε, είναι ιδέες οι οποίες ομοιάζουν ή συνάδουν με τη στρατηγική ασφαλείας ε, που παρουσίασε η κυρία Μογκερίνη. Σας είπα ότι η συνεργασία με τον ΝΑΤΟ είναι ζωτική σημασίας και το γνωρίζετε για ποιο λόγο. Όπως επίσης και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών. επειδή η εξωτερική και η εσωτερική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, τείνουν να συγχωνευθούν, θα έλεγα ότι και τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας θα πρέπει να συγχωνευτούν. Επομένως, πρέπει να υπάρχει ένα συνεχές ε, φάσμα δράσεων και μέσων για όλες τις περιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν. Και αυτά φυσικά θα πρέπει να ενδυναμώσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και να της δώσουν τη δυνατότητα να δράσει σε όλο το σπάσμα μέχρι του άρθρου ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν είναι μόνον καλοπιστικού χαρακτήρα αλλά το έχει ήδη επικαλεστεί η Γαλλία. Όσον αφορά την ε, κρίση ή τις κρίσεις, αυτό το οποίο ήθελα να αναφέρω σε αυτή την έκθεση είναι ότι πρέπει να ιεραρχήσουμε τις κρίσεις και τις σειράξεις τις οποίες θέλουμε να συμμετέχουμε και να έχουμε στην κορυφή της λίστας ε, κρίσεις οι οποίες επηρεάζουν άμεσα την ασφάλειά μας. Υπάρχουν κάποιες κρίσεις οι οποίες δεν είναι τόσο σημαντικές για την ασφάλειά μας. Ε, θα μπορούσαμε ίσως να δεχτούμε να, να συμμετέχουμε και σε αυτές, αλλά αυτές ε, οι δράσεις είναι ε, πιο πολύ για λόγους επίδειξης και δεν έχουν άμεση σχέση με την ασφάλειά μας. Θα πρέπει λοιπόν, θα υποχρεωθούμε μάλλον να ιεραρχήσουμε τις προτεραιότητές μας πρέπει να αναθεωρήσουμε το θέμα των μονάδων μάχης. Οι μονάδες μάχης πρέπει να γίνουν απαραίτητο εργαλείο, αποτελούν ε, ένα μέσο το βιτρίνα αυτή τη στιγμή, τις κοιτάμε, τις θαυμάζουμε, αλλά δεν έχουν ακόμα κινητοποιηθεί. Πρέπει επίσης να υπάρχει αυξημένη ε, ε, δυνατότητα να είμαστε πιο ε, ευέλικτοι και να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις μονάδες μάχης όσο καλύτερα μπορούμε. Όσον αφορά το θέμα της συνεργασίας με τον ΝΑΤΟ, οι δύο οργανισμοί δεν έχουν την πολυτέλεια να επαναλαμβάνουν τα ίδια πράγματα και αυτό το οποίο βλέπουμε είναι μια συμπληρωματικότητα. Ενώ το ΝΑΤΟ είναι σχεδιασμένο και εξοπλισμένο για να αντιμετωπίζει θέματα άμυνας και να εφαρμόσει συλλογική άμυνα, το άρθρο 5, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ε, σε θέση να αντιμετωπίσει προκλήσεις που αφορούν την εσωτερική ασφάλεια των κρατών μελών και ε, συμπεριλαμβανομένες και της αποτροπής που δεν καλύπτονται από το κεφάλαιο 5. Επομένως, από το άρθρο 5 υπάρχει μια λογική συμπληρωματικότητα μεταξύ των δύο οργανισμών και ε, η συγχώνευσή τους, ε, η συνεργασία τους μάλλον, θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε καλύτερα αυτές τις προκλήσεις. Ε, επικροτούμε την κοινή δήλωση που υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία και υποστηρίζουμε απόλυτα και τα περιθώρια συνεργασίας που αναφέρονται εκεί. Υπάρχει και ένα θέμα το οποίο πρέπει να εξετάσουμε. Δεν αναφέρεται στην έκθεση, αλλά θα πρέπει να το εξετάσουμε. Τώρα που η Βρετανία θα αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα παραμείνει μέλος του ΝΑΤΟ. Σχόλια εκτός μικροφώνου. Ε, όχι θα παραμείνουν, γιατί από τη μια υπάρχει λόγος για να συμμετέχουν με την άμυνα και την ασφάλεια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ταυτόχρονα η σχέση με το ΝΑΤΟ γίνεται ουσιαστική πλέον. Και εδώ γνωρίζετε πολύ καλά ότι περιμένουμε από τη Βρετανία να υποστηρίξει την Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέμα αυτό. Τώρα, υπάρχουν επίσης και εξελίξεις ε, στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, στην έρευνα για τη τεχνολογική βάση που αναφέρονται και αυτές στην έκθεση. Και ξεκινούμε λοιπόν από την εξή πραγματικότητα. Ο τομέας της αμυντικής βιομηχανίας στην Ευρώπη είναι κατακαιρματισμένος, αλλά αν θέλουμε να άρουμε αυτά τα προσκόμματα, πρέπει να υπάρχει κοινό ενδιαφέρον από όλα τα κράτη-μέλη. Δεν θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα αφορά λίγες χώρες ή λίγες επιχειρήσεις και όλοι οι υπόλοιποι θα πρέπει να ακολουθούν. Σε καμία περίπτωση αυτό δεν αποτελεί συνταγή επιτυχίας. Μια κοινή αγορά άμυνας, βεβαίως, αυτό είναι το επιθυμητό για πολλούς και διάφορους λόγους, δεν το αφισβητούμε αυτό, αλλά ταυτόχρονα θα θέλαμε αυτή η κοινή αγορά άμυνας να υποστηρίζει τις χώρες μέλη όταν υπάρχουν ε, συγκεκριμένες απειλές και προκλήσεις που αφορούν αυτά. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη, διότι θα πρέπει να απαντούν στα αιτήματα όλων. Λέμε και υποστηρίζουμε ε, πράγματα για την, ε, ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας, ο οποίος αποτελέσει τον πυλώνα για όλες αυτές τις προσπάθειες και φυσικά υποστηρίζουμε και τη σταδιακή συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ε, δραστηριότητες που αφορούν ε, στην άμυνα. Μέσω έρευνας, ε, σχεδιασμού, προγραμματισμού και υποστηρίζουμε και το πρόγραμμα δράσης για την άμυνα και την αμυντική βιομηχανία εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω ε, εκτεταμένης και πολύ καλά σχεδιασμένης έρευνας και ζητάμε και κατάλληλη χρηματοδότηση για το υπόλοιπο του πολιετές δημοσιονομικού πλαισίου, λαμβάνοντας υπόψη και ένα ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα στο επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Σε γενικές αδρές γραμμές αυτή είναι η εκθεσή μου. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από όσο γνωρίζω δεν βρίσκονται εδώ όλοι οι σκιώδεις εισηγητές. Ο κύριος Ντανζόν είναι σκιώδης εισηγητής για το ΕΛΚ. Αλλά νομίζω ότι ο κύριος Γκάλερ θα μιλήσει εκ μέρους του. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, ναι, ο κύριος Ντανζόν δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα και μου ζήτησε να παρουσιάσω τη θέση του. Ε, Ιωάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχέδιο. Είναι ένα πάρα πολύ καλό περιεκτικό σχέδιο έκθεσης και ο κύριος ε, Ντανζάν συμμερίζεται την προσέγγιση που ακολούθησε. Ασχολείται με τα ε, θέματα που είναι τρέχοντα αυτή τη στιγμή την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Ε, ζητάς μια αναθεώρηση και τη θεωρούμε αναγκαία δεδομένων των προκλήσεων στην ασφάλεια. Επίσης, στηρίζουμε αυτήν την διασύνδεση ανάμεσα στην εσωτερική και την εσωτερική ασφάλεια που τόνισες. Δεν μπορούμε να τις χωρίζουμε με τον παραδοσιακό τρόπο όπως κάναμε μέχρι τώρα. Διότι πλέον ο χαρακτήρας είναι διασυνοριακός και επιβάλλει καλύτερη συνεργασία, ανταλλαγή πληροφοριών και Επίσης, η... χρειάζεται καλό συντονισμό των φορέων εξωτερικής και εσωτερικής ασφάλειας. Χρειάζεται συνεργασία, λοιπόν. Επίσης, ο κύριος Νταντζάν θα ήθελε να τονίσει ότι στηρίζει την αναφορά στη... σε μια παγκόσμια στρατηγική και θεωρεί επίσης καλό πως ε, τονίζεται η αναγκαία συνεργασία με τον ΝΑΤΟ. Επίσης, θα ήθελα να προτείνει την συμπερίληψη της ε, συνεργασίας και με άλλους διεθνείς οργανισμούς για να τονιστεί αυτή η παγκόσμια διάσταση της συνεργασίας. Η αναθεώρηση επίσης των αποστολών και των επιχειρήσεων στα πλαίσια της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας θεωρεί ο κύριος Ντανζάν πως ε, είναι πολύ σημαντική. Γι' αυτό καλό είναι να τονιστούν τα πιο προβληματικά σημεία και θα υποβάλει τις σχετικές τροπολογίες. Επίσης, θα ήθελα να αναφερθεί και η ε, πρωτοβουλία CSBD. Αυτά λοιπόν μου έδωσε εντολή να αναφέρω ο κύριος Νταντζάν. Σε γενικές γραμμές θα ήθελα να πει πως ε, το σχέδιο έκθεσης είναι πολύ καλό και σίγουρα θα σας στήριξη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Τζέφρι Βανόρδεν έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ιωάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και δεδομένου του θέματος, πιστεύω πως η προσέγγιση που υιοθέτησε είναι αρκετά ε, λογική. Ιδιαίτερα μάλιστα εφόσον αναγνωρίζεις τη σημασία του ΝΑΤΟ. Στην έκθεσή σου διατυπώνεις το ερώτημα του ε, τι ακριβώς είναι η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Μέχρι τώρα έχουμε εστιάσει στη διαχείριση κρίσεων και παρόμοιες ε, ε, πτυχές. Όμως η πολιτική αυτή έχει να κάνει και με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Και αυτό πιστεύω πως είναι και η κινητήριος δύναμη. Και εάν λείπει αυτό, τότε η λογική της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας διαλύεται. Επίσης η πολιτική αυτή είναι κάτι που διχάζει. Διχάζει δηλαδή με την έννοια ότι προσπαθεί να δημιουργήσει ένα τεχνητό ευρωπαϊκό μπλοκ το οποίο θα είναι ξεχωριστό από τις ΗΠΑ ή από οποιαδήποτε άλλη διατλαντική συμμαχία. Και πιστεύω πως αυτό είναι και το αγγενές λάθος ε, εδώ, διότι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η ασφάλεια και η άμυνα θα είναι μόνον αξιόπιστε εάν διασφαλίσουμε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε θα συνεχίσουν να ε, συμπεριλαμβάνονται 100% στην ε, πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών. Και αυτό είναι και ο ρόλος του ΝΑΤΟ στην ουσία. Δεν χρειάζεται βέβαια να ακούσετε και από μένα το πόσο σημαντικό είναι το ΝΑΤΟ, αλλά από τη μία ακούγονται όλα αυτά τα ωραία λόγια και από την άλλη προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια ξεχωριστή οντότητα, στόχος της οποίας είναι στην ουσία να υπονομεύσει το ρόλο του ΝΑΤΟ. Χρειάζεται λοιπόν να ε, αναζωογονηθεί η ε, συμμαχία και να δηλωθεί ξανά ξεκάθαρα η δέσμευση της Ευρώπης σε αυτή. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση τόσο για τις στρατιωτικές δαπάνες όσο και για την συμμετοχή σε στρατιωτικές επιχειρήσεις όπου εκείνο χρειάζεται. Αυτό βέβαια δεν θα γίνει μέσω ε, της ε, κοινή ε, πολιτικής ασφάλειας και άμυνα. και επίσης ε, νομίζω πω ε, και σε πρόσφατες συζητήσει που είχαμε για την Ευρωπόλ ακούστηκε ο τελικός στόχος, η δημιουργία δηλαδή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνα. Δεν είμαι σίγουρος για το σκοπό όλων αυτών και δεν είμαι σίγουρος για το πότε οι πολίτες της Ευρώπης θα καταλάβουν ότι πηγαίνουμε προς τη λάθος κατεύθυνση. Δεν είναι αυτό που θέλουν οι πολίτες μας. Γι' αυτό θεωρώ ότι οι συζητήσεις σε επιτροπές όπως αυτή δεν είναι αντιπροσωπευτικές του αισθήματος που υπάρχει ανάμεσα στους πολίτες των ε, κρατών μελών. Χρειάζεται μια ισχυρή άμυνα μέσω του ΝΑΤΟ που θα διασφαλίζεται και από τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης, αναφέρεστε στην ανάγκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμμετέχει σε ε, προσπάθειες ε, ανατροπής ανατροπών. Βλέπουμε προς τις πρόσφατες εξελίξεις με, τους, ε, με τις υβριδικές απειλές, με τη συμμετοχή της Ρωσίας. Όμως η ανατροπή δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό. Ιστορικά η ανατροπή ήρθε μέσω του κομμουνισμού και μέσω των πολιτών της ε, ίδιας μας της χώρας οι οποίοι είχαν τέτοιες πεπιθήσεις. Στην ουσία αυτό που βλέπουμε τώρα είναι πως υπάρχει μία ε, νέα εμφάνιση αυτών των τάσεων. Βλέπουμε ότι η ηγεσία του Εργατικού Κόμματος, ε, για παράδειγμα, στη χώρα μου έχει πέσει θύμα αυτών που θεωρούσαμε ε, τε, ε, παλιές ξεχασμένες ιστορίες. Γι' αυτό λοιπόν ε, ας μην ξεχνάμε ότι όταν γίνεται λόγος για ανατροπή πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και αυτού του είδους οι ανατροπές. Τώρα στη Ρωσία αναδύεται ξανά ο μαρξισμός και ο λεμισμός, ε, στη Μέση Ανατολή τζιχαντισμός, ο οποίος δεν παραμένει μόνο εκεί αλλά έρχεται και ε, στα σπίτια μας και αυτή είναι η ανατροπή για την οποία μιλώ. Και το τελευταίο που χρειαζόμαστε είναι η ανάμειξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πολιτική εσωτερικής ασφάλειας στις χώρες μας. Τώρα, φυσικά και θέλουμε στενή συνεργασία ανάμεσα στις υπηρεσίες ε, ε, πληροφοριών και ασφάλειας. Όμως, ας μην προχωρήσουμε υπερβολικά πολύ. Ας μην ε, αναμίξουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ. Μάλιστα υπήρξαν και πολλές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ, οι οποίες είναι αντιπαραγωγικές. Έτσι αποδείχθηκε. Και μάλιστα υπονόμευσαν το διεθνές δίκαιο για το άσυλο, για παράδειγμα. Βλέπουμε λοιπόν ότι με την συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα προβλήματα επιδεινώθηκαν. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ πως ε, βαδίζουμε προς τη λάθος κατεύθυνση. Τώρα, παρά το γεγονός ότι επικροτούμε την αναφορά στο ΝΑΤΟ, όλες οι υπόλοιπες αναφορές στην δημιουργία τεχνητά μίας ε, ευρωπαϊκής υπηρεσίας, η οποία θα εμπλέκεται στη, στα θέματα ασφαλείας των χωρών μας, είναι κάτι με το οποίο δεν συμφωνούμε. Ευχαριστώ πολύ. Σκιώδης εισηγητής για τους φιλελεύθερους είναι ο κύριος Ράντος, αλλά... Ο κύριος Αυστρεβίτσιος θα μιλήσει εκ μέρους του, διότι απουσιάζει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για μία περιεκτικότατη έκθεση σχετικά με την πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους του συναδέλφου κυρίου Ράντος, ο οποίος ε, απουσιάζει λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων στη χώρα του. Μαντέψτε για ποια χώρα μιλάω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα αντιμετωπίζει βαθιές αλλαγές στο τοπίο ασφάλειας. Οι κοινωνικές, οικονομικές, οι τεχνολογικές και οι γεωπολιτικές τάσεις συνδέονται άμεσα. Το τοπίο λοιπόν αλλάζει συνεχόμενα και αλλάζουν και οι προκλήσεις. Η πολιτική μας ομάδα λοιπόν θεωρεί ότι χρειάζεται ενότητα για να απαντήσουμε έγκαιρα και κατάλληλα. Γι' αυτό λοιπόν στηρίζουμε την θεμελιώδη αναθεώρηση της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, διότι θεωρούμε ότι όπως αναφέρατε στα πλαίσια της νέας στρατηγικής ασφάλειας, υπάρχει μεγάλη ανάγκη για συνεργασία και συντονισμό των πολιτικών ασφαλείας και άμυνας και θεωρούμε πως οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ενισχύσουν τη συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη, θα ενισχύσουν τη λειτουργία των Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών ε, Πληροφοριών και θα οδηγήσουν στην δημιουργία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας. Ε, Επίση, η περαιτέρω ολοκλήρωση των ε, υπηρεσιών ασφάλειας και άμυνας είναι κάτι το οποίο θεωρούμε πως είναι θετικό και θα ενισχύσει την ανθεκτικότητα και την αποτελεσματικότητα της Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Λόζιν έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Να σας δώσω και λίγο χρόνο να φορέσετε τα ακουστικά σας. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν κύριε Πάσκου. Δεν θα σας εκπλήξει φαντάζομαι το ότι πρέπει να πω εκ μέρους της πολιτικής μας ομάδας ότι έχουμε θεμελιώδεις διαφορές με τη... τα όσα γράφετε στην έκθεσή σας. Έχουμε μια διαφορετική κατανόηση της κατάστασης και εσείς κύριε Πάσκου μιλάτε για ανάλυση κρίσεων και για την στρατηγική που θα ακολουθήσει για τη διαχείριση αυτών των κρίσεων. Θα ήθελα να σταθώ σε ορισμένα πράγματα. Για παράδειγμα, για μας πάρα πολύ σημαντικό είναι να ε, δοθεί ένα σαφής σε της τρομοκρατίες και του πολέμου. Τι εννοούμε με το ένα, τι εννοούμε με το άλλο. Κάτι το οποίο τελευταία ε, Οι δύο ορισμοί συγχαίονται. Η τρομοκρατία τον τελευταίο καιρό αντιμετωπίζεται από την αστυνομία και πιστεύω πως χρειάζεται να συζητηθεί ε, για να συζητηθεί το αν χρειάζεται διαφορετική κατάρτιση, διαφορετικός εξοπλισμός από ε, την αστυνομία για την αντιμετώπιση τέτοιων ε, κρουσμάτων ε, τρομοκρατίας. Επίσης, θεωρώ εξίσου προβληματικό τον ορισμό του πολέμου και το πώς αυτό συνδέεται με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις όλα αυτά, ξέρετε, έχουν συνέπειες. Συνέπειες που είναι και συνταγματικές και για τα κράτη-μέλη και για τα συντάγματα αυτών. Συνέπειες οι οποίες μάλιστα είναι ευρύτατες και συνέπειες οι οποίες είναι πολύ σημαντικές για τη δημοκρατία. Και θεωρώ πως θα ήταν ολέθριο εάν η δημοκρατία μας ε, υπονομευθεί από τη δημιουργία τέτοιων οργανισμών οι οποίοι είναι αντίθετη στην δημοκρατία, στις αρχές της και στον δημοκρατικό έλεγχο. Αυτό λοιπόν ε, θεωρώ πως θα γίνει εάν ε, ε, ενωθεί η εσωτερική και η εξωτερική άμυνα και προστασία. Τώρα, θα σταθώ λίγο στις τρομοκρατικές απειλές, στην πρόληψη και στα αίτια. Πιστεύω πως η πολιτική θα έκανε λάθος εάν θωράκιζε ε, ακόμα περισσότερο τον εαυτό της, εάν γίνονταν ακόμα περισσότερες επενδύσεις στην άμυνα. Από ποια κονδύλια, από ποιον προϋπολογισμό. Υπάρχουν άλλα προβλήματα, υπάρχουν οι κοινωνικές ανισότητες, η καταπολέμηση της φτώχειας με τα οποία πρέπει να ασχοληθούμε. Και έτσι θεωρώ πως, ε, είναι, πως γίνεται η καλύτερη δυνατή πρόληψη της τρομοκρατίας. Κύριε Πάσκου, επίσης αναφέρεστε με πολύ θετικά σχόλια στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για παράδειγμα, αναφέρεστε στην εφαρμογή ε, για στην, εφαρμο... Ε, χρήση μάλλον κονδυλίων για την άμυνα που θα προέρχονται από άλλους ε, τομείς του προϋπολογισμού. Βλέπω πως ε, προσανατολισόμαστε όλο και περισσότερο προς ε, έναν στρατιωτικό χαρακτήρα της ε, πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Και θεωρώ πως οι αντιδράσεις του κοινού θα είναι πάρα πολύ έντονες, ιδιαίτερα μάλιστα όταν ε, κονδύλια τα οποία προορίζονται για ανθρωπιστική βοήθεια δοθούν στην ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων. Επίσης, πρέπει να μιλήσουμε για την μετανάστευση, πρέπει να μιλήσουμε για τους πρόσφυγες και για τις αιτίε που δημιουργούν προσφυγικές ροές. Οι αιτίε που δημιουργούν λοιπόν ε, προσφυγικές ροές συνδέονται επίσης άμεσα με τους ελέγχους στα σύνορα. Δεν μπορούμε να κάνουμε το ένα χωρί το άλλο. Δεν μπορούμε να διενεργούμε απλά έλεγχου στα σύνορα, να τα κλείνουμε χωρί να προσπαθούμε πιο πριν να καταπολεμήσουμε τα αίτια τη φτώχεια, τα αίτια που δημιουργούν πρόσφυγε. Γι' αυτό λοιπόν και για όλα αυτά που είπα, έχουμε έντονα επικριτική στάση απέναντι στην έκθεσή σα. Θα την καταψηφίσουμε, θα υποβάλουμε μία ε, έκθεση μειοψηφίας και επίσης σχετικές τροπολογίες στην έκθεσή σας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Βαλέρο. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ με τον κύριο Πάσκου. Όντω υπάρχουν νέε προκλήσει. Όμω, μέχρι εκεί τα σημεία συμφωνία μα. Νομίζω ότι έχουμε πολύ διαφορετικέ απόψει ω προ το πώ μπορούμε να διαμορφώσουμε την ασφάλεια για του πολίτε μα. Ο κύριο Πάσκου έχει έναν πιο στρατιωτικό τρόπο αντίληψη, εγώ ε, πιο πολιτικό. Είπε ο κ. Πάσκου ότι αποτελεί ένα μέσο διαχείρισης εκρίσεων. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε πολύ περισσότερο και στα μέτρα πολιτικής προστασίας, αποτροπής ε, συγκρούσεων και το καθεξής και να μην στεκόμαστε μόνο στην στρατιωτική διάσταση. Και συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Λέσσινγκ για την τρομοκρατία και τον πόλεμο αρχίζουμε να αποκαλούμε αυτή την κατάσταση ε, ανταρτοπόλεμο, τότε είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε στρατιωτικά. Προς το παρόν έχουμε μια αστυνομική αστυνομική αντιμετώπιση και πολύ ορθά, γιατί ε, είναι η αστυνομία που θα πρέπει να το αντιμετωπίσει. Όταν όμως μιλούμε για ανταρτοπόλεμο, ε, τότε έχουμε τε, τελείως διαφορετικό σημείο εστίασης. Ο κύριος Βανόρντεν επίσης ε, αναφέρθηκε στο ΝΑΤΟ. Για παράδειγμα, στην πατρίδα μου δεν περιμένει κανείς από το ΝΑΤΟ ή από τις ΗΠΑ να μας υπερασπιστεί. Δεν θέλουν καν να συμμετέχει η χώρα μας ε, στο ΝΑΤΟ και μάλιστα πολλές φορές αντιτίθεται και σε στερεωτικές ε, επιχειρήσεις και και ασκήσεις μάλλον. Είναι σημαντικό να το έχουμε αυτό κατά νου όταν συζητούμε τέτοια ζητήματα κοινή ασφάλειας, κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνα, ότι δεν θέλουν όλε οι χώρε αυτή ακριβώ τη συμμετοχή και ενίσχυση τη συνεργασία. Γιατί σε όλα τα κείμενά μα συνήθω υπάρχει μια μεγάλη ε, συγχαίωμα αρκετά την Ευρωπαϊκή Ένωση με το ΝΑΤΟ. Εδώ έχουμε και το άρθρο 14 για παράδειγμα που εσεί, κύριε Πάσκου χαιρετίζετε την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ανέφερε η κυρία Λόζινγκ Πραγματικά όμως εγώ την καταδικάζω στα νερά γιατί προσπαθούμε να αντλήσουμε κονδύλια από την ανάπτυξη και να τα δαπανίσουμε στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Αυτή τη συζήτηση κάναμε και χθες στην Πρατισλάβα ή χθες ή προχθές. Όταν μιλούμε για χώρες που ακόμα δεν φτάνουν τον ε, στόχο του 0,7 για την ανάπτυξη, και εμείς μάλιστα θέλουμε να περιορίσουμε αυτά τα κονδύλια για να τα δαπανίσουμε σε στρατιωτικέ επιχειρήσεις, ακόμα και αν δεν είναι άμεση η ενίσχυση, για παράδειγμα, των στρατιωτικών εξοπλισμών, ακόμα και εμέσως πρόκειται για αναπτυξιακή βοήθεια και αντί να χρησιμοποιείται για την διαμονή, την παιδεία, την υγειονομική περίθαλψη και για όλα αυτά τα πράγματα που μπορούν να αλλάξουν πραγματικά τις ζωές των ανθρώπων και να διαμορφώσουν ένα πλαίσιο ασφάλειας στις πατρίδες τους, θα τα πανούμε αλλιώ. Γιατί όταν έχουμε μια προηγμένη χώρα είναι και πολύ πιο ασφαλής, αλλά και λιγότερο στρατητικοποιημένη. Νομίζω ότι η συζήτηση αυτή θα συνεχιστεί με μεγάλο ενδιαφέρον και σίγουρα δεν θα συμφωνήσουμε σε μεγάλο βαθμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Σκελάμ. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ στηρίζω την πρωτοβουλία του συναδέλφου κ. Πάσκου και την προσέγγισή του, γιατί εδώ μας παρουσιάζει μία έκθεση που περιλαμβάνει και μία διάγνωση η διεθνής κατάσταση προς την ασφάλεια είναι περίπλοκη, επιδεινώνεται και δεν υπάρχει μια πραγματικά συντονισμένη και αποτελεσματική συλλογική αντιμετώπιση. Αυτό είναι το κύριο πρόβλημα. Έχουμε πολλές διακηρύξεις, δηλώσεις, προγράμματα, καλές προθέσεις. Όμως υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ των διακηρύξεων αυτών και της υλοποίησής τους. Και καθυστερούμε να αντιδράσουμε στις ε, πλέον περίπλοκες και σύνθετες κρίσεις. Γι' αυτό και ο τίτλος του εγγράφου μιλά για υλοποίηση. Και νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα της αλήθειας για μας. Θα σταθούμε σε ακόμα μία τέτοια σύνθετη διακήρυξη ή θα προχωρήσουμε σε κάτι πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου. Να μετατοπιστεί το σημείο έμφαση από την διαχείριση κρίσεων, που βεβαίω είναι κάτι το οποίο κάνουμε, στην πρόληψη κρίσεων και επίλυση κρίσεων, όπως αναφέρεται. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλη λύση στη σημερινή κατάσταση. Αν θέλουμε να την αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα. Άλλος συνάδελφος ανέφερε την σύνδεση μεταξύ της ε, εσωτερικής και εξωτερικής κατάστασης προς την ασφάλεια είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει, όμως ε, από πρακτικής άποψης δεν είμαστε έτοιμοι να το πράξουμε. Παρατήρησα και την προσέγγιση σας ως προς τη χρήση των ε, μέσων διατήρησης ε, της ειρήνης. Δεν θέλουμε να αμελήσουμε, να παραλείψουμε ε, το πεδίο εφαρμογή αυτών των μέσων, όμως θα πρέπει να τα διευρύνουμε για να ανταποκριθούμε ε, στις έντονες αυτές ε, οξύες κρίσεις, όπου η στρατητική μας στήριξη σε συγκεκριμένους φορείς θα βοηθούσε για να έχουμε και περισσότερες δυνατότητες σταθεροποίησης της κατάστασης. Εδώ το βασικό στοιχείο δεν είναι πώς η δική μας κοινή γνώμη θα αντιδρούσε, αλλά πώς θα μπορούσαμε να επιλύσουμε την κρίση. Όταν βρισκόμαστε με δεμένα τα χέρια ουσιαστικά, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε, να το συζητήσουμε επισταμένως και να αποφασίσουμε. Τέλος, Μιλήσατε και σε μια τεχνολογική και βιομηχανική ε, βάση, αμυντική βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα πρέπει να ενισχυθεί. Είναι θεμελιώδες στοιχείο για μια αποτελεσματική κοινή πολιτική ε, ασφαλεια και άμυνας. Και βέβαια η συμπληρωματικότητα ως προς το ΝΑΤΟ είναι προφανέστατη. Δεν μπορούμε να δημορφώσουμε μια ξεχωριστή ε, πολιτική ασφαλείας και άμυνας πρέπει να συνεργαστούμε με το ΝΑΤΟ. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε αλληλεπικαλύψεις ως προς τις ε, προσπάθειές μας ε, και την αξιοποίηση των κονδυλίων. Βεβαίως, οι προτεραιότητες ως προς το ΝΑΤΟ θα πρέπει να τηρηθούν. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Ασενκάν. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ ξεκινώντας να πω ότι χαιρετίζω την έκθεση του συναδέλφου Πάσκου και τα όσα προανέφερε. Σε αδρές γραμμές πρόκειται για μια καλή προσέγγιση. Αναμφίβολα, κατά τη γνώμη μου, διερχόμαστε δύσκολες ε, περιόδους, δύσκολους καιρούς, με πολλές προκλήσεις και παλαιότερες και νεότερες. Πολλές από αυτές είναι σύνθετες και όντως χρειαζόμαστε μια αποτελεσματική απάντησε και ανταπόκριση. Η Συρία θεωρώ ότι είναι ένα καλό παράδειγμα, όπου αποτύχαμε να ανταποκριθούμε γρήγορα και αποτελεσματικά και αυτό οδήγησε σε τεράστια προβλήματα. Και νομίζω ότι αυτό το παράδειγμα καταδεικνύει ότι όταν όταν δεν παρεμβαίνουμε, ακόμα και το πρόβλημα είναι μακριά από εμά, κάποια στιγμή φτάνει και στην πόρτα μα. Η τρομοκρατία είναι ακόμα ένα τέτοιο ζήτημα. Υπάρχει ένα σύνθετο ε, ιστορικό υπόβαθρο βεβαίω, αλλά ξέρουμε ότι πλέον αυτό το ζήτημα έχει γίνει και δικό μα πρόβλημα. Και θα πρέπει να εργαστούμε συλλογικά για να το αντιμετωπίσουμε. Για την κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνα, θεωρώ και πάλι ότι όσο περισσότερο εξετάζουμε δυσκολίε και προκλήσει που υφίστανται, τόσο περισσότερο βλέπουμε πόσο λεπτό είναι το ζήτημα και νευραλική σημασία. Πρέπει ακριβώς να συνεργαστούμε. Και εγώ προέρχομαι από την ίδια χώρα με τον ε, Τζέφρι Βαν Όρντεν. Αλλά θα σας πω το εξής. Είναι κάτι το απαραίτητο. Δεν πρόκειται ε, για κάτι που υποκαθιστά το ΝΑΤΟ, αλλά το συμπληρώνει θεωρώ ότι ακόμα και η Βρετανική κυβέρνηση στηρίζει ε, την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Ε, είναι διατεθειμένοι να συνεργαστούν με του υπολείπου και οτιδήποτε και αν συμβεί κατόπιν του δημοψηφίσματο, θα υπάρξει συνεργασία σε αυτόν τον τομέα. Το κατανοούν και εκείνοι. Ήθελα επίσης να σταθώ σε κάτι το οποίο ανέφερε ο Τζέφρι στο κόμμα των εργατικών. Εγώ είμαι μέλο των εργατικών και χαίρομαι που είχαμε το μεγαλύτερο πολιτικό κόμμα στην ε, Ευρώπη. Δεν θεωρώ ότι οι κομμουνιστές αναλαμβάνουν ε, την ηγεσία ε, των εργατικών. Γι' αυτό θεώρησα μου να αμφισβητήσω αυτή την δήλωση. Είναι πολύ καλή η προσέγγιση του εισηγητή. Θα κάνω κι εγώ κάποιες επισημάνσεις, όμως νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή αφετηρία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι αυτό ήταν το τελευταίο αίτημα. Να δώσω το λόγο στον κύριο Πάσκου για να συνοψίσει. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ όλους που ασχοληθήκατε με το θέμα αυτό στις διακοπές και διαβάσατε την έκθεση και Γι' αυτό ακριβώ και κάνετε και πολύ σημαντικές παρατηρήσεις. Κάποιες ε, οδεύουν προς την ίδια κατεύθυνση με τη φιλοσοφία τη έκθεσης, κάποιες άλλες όχι, αλλά είναι εξίσου σημαντικές, ε, διότι οι συνάδελφοί μας εξετάζουν πολύ σοβαρά το θέμα αυτό και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Συμφωνώ με τον κύριο Γκάλερ και με τον Αρνό αν θέλουμε να αλλάξουμε σημείο και να περάσουμε από τι επιχειρήσεις σε πραγματική πολιτική ασφάλεια και άμυνα Να πω εδώ ότι δεν αναφέρθηκα πολύ στις επιχειρήσεις εν εξελίξη και δεν ε, αναφέρθηκα και πολύ στη σχέση με άλλους διεθνείς οργανισμούς που όπως γνωρίζετε είναι επίσης παρόντες στις περιοχές τις οποίες έχουμε επιχειρήσεις. Το δέχομαι φυσικά αυτό, σαφέστατα και θα υπάρξουν τροπολογίες. Θα τις επαστώ αυτές τις τροπολογίες και θα τις συμπεριλάβω στην έκθεση για να συμπληρώσω το σχετικό κεφάλαιο. Για τα όσα είπε ο Τζόφρι. Ε, δεν τα ακούω και πρώτη φορά, τα συζητάμε και δημοσίως και ιδιωτικώς εδώ και χρόνια. Αν όμως συζητάμε το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένε Πολιτείες, το 50% ε, των μελλοντικών εξελίξεων ε, έρχεται να αρνηθεί αυτά τα οποία θεωρείται εσείς δεδομένα ο ένας υποψήφιος λέει αυτά που λέτε κι εσείς. Θα ελέγξει κατά πόσο οι σύμμαχοι έχουν ε, πληρώσει αυτό που τους αναλογεί και κατά αν και εφόσον το έχουν πληρώσει τότε θα τους υποστηρίξω Τους άλλους θα τους πούμε συγγνώμη, ευχαριστούμε πολύ, κοιτάξτε κάπου αλλού. Αυτό δεν είναι ε, μια ωραία εικόνα για το μέλλον. Δεν μπορείς λοιπόν Τζέφρι να μου λες ότι δεν μπορούμε να τα λάβουμε σοβαρά υπόψη και δεν χρειάζεται να τα λάβουμε υπόψη. Εάν όντω συμβεί κάτι τέτοιο, εμείς που βρισκόμαστε, η Ευρώπη που βρίσκεται. Θα βασιζόμαστε ακόμα σε ένα ΝΑΤΟ το οποίο δεν θα λειτουργεί. Υπάρχει πρόβλημα λοιπόν και νομίζω ότι γνωρίζετε ότι και οι Αμερικανοί και αν ε, σκεφτώ και το Πανέτα και το Gates, και αυτοί είπανε κάντε περισσότερα για το θέμα αυτό να βρούμε μια μέση λύση. Και αυτό το οποίο κάνουμε είναι να προετοιμαστούμε για ένα τόσο ζωφερό μέλλον και ταυτόχρονα να, να προσπαθούμε να απαντήσουμε και στο αίτημα των συμμάχων μας. Καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να υπάρξει επιμερισμό του βάρου και το κάνουμε αυτό και στο ΝΑΤΟ. Το βλέπετε ότι υπάρχουν χώρε οι οποίε προσπαθούν να επιτύχουν αυτό το 2% και αυξάνουν τι δαπάνε του. Όταν αναφέρθηκα σε αυτό ε, και ε, ε, επεσήμανα ότι είναι συμπληρωματικός ο ρόλος και ότι δεν θέλουμε εμείς να αντικαταστήσουμε το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ δεν απαντά στις ίδιες προκλήσεις με τις οποίες είναι εξοπλισμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση να απαντήσει. Παραδείγματος χάρη, εγώ δεν σας είπα την ανατροπή. Εγώ την αντιλαμβάνομαι με τεχνικούς άρους. Είναι ένα προηγούμενο επίθεσης ε, στην κοινωνική δομή μιας χώρας. Αυτή είναι η ανατροπή. Δεν έχει σχέση αν έρχεται από τους κομμουνιστές ή από το Ισλαμικό κράτος. Από τεχνική σκοπιά αυτό είναι αποδυναμώνω τη χώρα στόχο μέσω υπονόμευσης και ανατροπής. Και το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να αποτελέσει πρόληψη στην ανατροπή. Και αν δείτε την ιστορία του ψυχρού πολέμου και την κορύφωσή του, οι Ηνωμένε Πολιτείε ήταν γεμάτες σοβιετικούς ε, κατασκόπους, σαμποτέρ και και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστείτε. Ανεξάρτητα λοιπόν από το άρθρο 5, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Και εδώ η παρατήρησή μου είναι ότι θα θέλαμε να ολοκληρώσουμε, να οικοδομήσουμε βάσει αυτών που έχουμε. Έχουμε για παράδειγμα αστυνομική συνεργασία μεταξύ διαφόρων οργανισμών. Έχουμε υπηρεσίε οι οποίε μαζεύουν του πάντε γύρω από ένα τραπέζι. Αυτά πρέπει να έχουμε κατά νου. Όχι να δημιουργήσουμε μια άλλη δομή στην οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπαίνει στα σπίτια μα να δει ε, αν είναι ασφαλή. χρησιμοποιούμε αυτά τα οποία διαθέτουμε ήδη, τα οποία τα έχουν δεχτεί άλλες χώρες, γιατί αλλιώς δεν θα τα είχαμε. Παραδείγματο χάρη, η ανατροπή και η υπονόμευση με τεχνικούς όρους και όχι με ιδεολογικούς όρους, γιατί αν αναφέρομαι σε ιδεολογικό πλαίσιο και σκέφτομαι μόνο στον κομμουνισμό, ε, τότε δεν υπάρχει λόγος να κάνει η Ρωσία αυτά που κάνει, γιατί δεν είναι πια κομμουνιστές. Και πριν από τον κομμουνισμό πάλι Ρώσοι ήτανε. Και πάλι τα αυτά έκαναν. Νομίζω ότι γνωρίζετε ότι το να προσεγγίσει κάποιος τεχνικά το ζήτημα είναι μάλλον ο μόνος τρόπος να μπορέσουμε ε, να παίζουμε επίσης όρις ε, στο θέμα αυτό. Κυρία Λούιζινγκ. Και εσείς κυρία Βαλέρο, μας λέτε ότι θέλουμε να πάρουμε λεφτά από την ανάπτυξη και να τα πάμε στην άμυνα. Ό,τι συνέβη, συνέβη με τα χρήματα για την ανάπτυξη που περιλαμβάνονταν ήδη στον προπολογισμό. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι κατά πόσον δεν επιτρέπουμε την επίτευξη αυτών των στόχων, διότι υπήρχαν αυτοί οι στόχοι ήδη Προσπαθήσαμε να του επιτύχουμε και ξαφνικά διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν ένα σωρό κρίσεις γύρω μας. Και τώρα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις κρίσεις και συμφωνώ μαζί σα. Οι πολίτες ε, θέλουν καλύτερα σχολεία για τα παιδιά τους, μια καλύτερη ζωή, θέσεις εργασίας. Αλλά άμα δεν μπορούν να βγουν από το σπίτι τους γιατί κάποιο πυροβολεί στη γωνία του δρόμου, ε, η αστυνομία και οι ενόπλες δυνάμεις, γιατί όλοι χρησιμοποιούν το στρατό Χωρί καμία φιλοσοφία επ' αυτού, διότι ο στρατό είναι αυτός ο οποίο είναι εξοπλισμένο να αντιμετωπίσει τη σοβαρότητα τη κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι πολίτε. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν με το θέμα αυτό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η συνοριοφυλακή ελέγχει την πραγματικότητα. Προσπαθεί να βρει μια λύση για να μπορέσει να ελέγξει ένα φαινόμενο το οποίο είναι πάρα πολύ αρνητικό ή μάλλον πάρα πολύ δύσκολο για μας. Και αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να, να φροντίσω. Αλλιώς θα δω στη συνέχεια τι θα κάνω με την ανάπτυξη εν γέννη. Και υπάρχει και κάτι ακόμα και σε τέτοιο στρατηγικό επίπεδο. Δεν μπορεί κάποιος να έχει ανάπτυξη εάν δεν έχει ασφάλεια. Και έρχομαι στο γιατί υποστηρίζω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να χρησιμοποιήσουμε τμήμα των κονδυλίων από το μέσο για αυτά τα πράγματα. Διότι ιδάλλως πρόκειται για λεφτά τα οποία τα πετάμε από το παράθυρο. Τους δίνουμε κάτι, τους οργανώνουμε λίγο, αλλά όταν χρειαστούν τα μέσα για να εφαρμόσουμε αυτά τα οποία τους διδάξαμε να κάνουν, δεν μπορούμε εμείς να τους δώσουμε τα μέσα και επομένω τα χρήματα τα οποία επενδύσαμε μέχρι εκείνη τη στιγμή πάνε από το παράθυρο και οι συγκρούσεις και οι σειράξεις συνεχίζονται. Δεν μπορούμε στην πραγματικότητα να επιλύσουμε τα προβλήματα. Γι' αυτό ακριβώ και είπα ότι επειδή έχω δει αυτές τις αποστολές, στον Ήγηρα, στο μαλί και διαμαρτύρονται ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Λένε δώστε μας και κάτι, να μην μας λέτε απλώς ότι να κάνεις αυτό και αυτό και εκείνο, και όταν ζητάμε για τα μέσα τους λέμε «Α, μέσα δεν μπορούμε να σας δώσουμε». Εκεί έγκυται το πρόβλημα. Εσείς δεν το λέτε ανταρτοπόλεμο γιατί δεν σας αρέσει. Πώς θα το βαφτίσετε. Όπως και να το βαφτίσατε, το γεγονός ότι πυροβολούν πολίτες στους ευρωπαϊκούς δρόμους ή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ε, εκρήγνιδες στους ευρωπαϊκούς δρόμους είναι πάρα πολύ σημαντικό και σοβαρό. Γι' αυτό και ακριβώς η ασφάλεια βρίσκεται στο επίκεντρο Τη ε, ανησυχία των Ευρωπαίων πολιτών. Αλλιώ δεν θα ήμασταν εκεί που είμαστε. Ακόμα θα περιμέναμε να γίνει ένα συμβούλιο σε δύο-τρία χρόνια να συζητήσει κατά πόσον, εάν και πόσον το επιτρέπει η μερίσια διάταξη, θα συζητηθεί κάτι για την άμυνα. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή είναι η ανησυχία των πολιτών. Οι ανησυχίε των πολιτών είναι πραγματικέ και οι πολιτικοί και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα προσπαθούν να απαντήσουν σε αυτέ. Ιδάλω, εάν και αυτή τη στιγμή εθελοτυφλούν, σημαίνει ότι χάνουμε την τελευταία μας ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε αυτά τα πράγματα. Αλλιώς θα μας περικυκλώσουν και δεν θα μπορούμε να αναπνεύσουμε εάν τους παραμολύσουμε, τους αγνοήσουμε και τους αφήσουμε στον ιδεώδη κόσμο της ανάπτυξης και της ευτυχίας για όλους. Ναι, αυτό θέλουμε. Και ας ελπίσουμε ότι θα τα καταφέρουμε. Λοιπόν, αυτά ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βανόρτερν ζήτησε εκ νέου το λόγο. Παρακαλώ. Ε, πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε. Όποιος ε, και αν είναι ο επόμενος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών σίγουρα θα ζητήσει και η Ευρώπη και οι άλλοι σύμμαχοι να κάνουν περισσότερα. Ε, εγώ θεωρώ ότι η απάντηση σε αυτό δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας. Κάτι άλλο. Αναφέρατε αυτήν την υπηρεσία πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και ταυτόχρονα μιλήσατε για ανατροπή. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ μία πιο ευάλωτη ευρωπαϊκή υπηρεσία, ευάλωτη στην ε, δίσδυση... Ε, κατασκόπων κτλ. από ότι την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Πληροφοριών. Αυτό είναι κάτι που για να γίνει σωστά προϋποθέτει ανταλλαγή πληροφοριών, προϋποθέτει καλή συνεργασία και τον απόλυτο έλεγχο του τι γίνεται. Και το τελευταίο πράγμα που χρειαζόμαστε είναι άλλη μία ευρωπαϊκή υπηρεσία, άλλον έναν ευρωπαϊκό οργανισμό, ο οποίος να έχει ε, στη διάθεσή του απόλυτες πληροφορίες. Συνάδελφοι, λέει η Πρόεδρος, ε, ξέρω πως ζητάτε το λόγο, όμως έχουν ήδη φτάσει οι προσκεκλημένοι μας, γι' αυτό θα σας παρακαλέσω να είστε σύντομοι. Ο κύριος Γκάλερ, σας ευχαριστώ. Συμφωνώ με το ότι η, Ευρωπαϊκός, ε, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Πληροφοριών δεν πρέπει να μας απασχολεί, δεν πρέπει να το συζητάμε καν. Όμως θεωρώ ότι δεδομένης της ανεπάρκειας που υπάρχει στις αμυντικές δαπάνες. Ίσως η χώρα σας, δεν ξέρω, είναι τόσο τέλεια, μπορεί να τα κάνει όλα μόνη της. Όμως υπάρχουν άλλες χώρες οι οποίες συνεργάζονται ε, καλύτερα. Και είναι πρακτικά τα ωφέλη της συνεργασίας. Αυξάνεται η διαλειτουργικότητα, τα αποτελέσματα είναι ε, καλύτερα πιο γρήγορα. Γι' αυτό θεωρώ πως είμαστε σε καλό δρόμο εάν συνεργαζόμαστε και συνεχίσουμε τη συνεργασία, διότι η ευρωπαϊκή ενιαία αγορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και προϊόντα τα οποία δεν είναι ε, μόνο ε, οικονομικά, αλλά μεταφράζονται και σε ικανότητες. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Βαλέρο έχει το λόγο. Ε, θα ήθελα και εγώ να σχολιάσω αυτό που είπατε για την ανάπτυξη. Εάν χρησιμοποιηθούν κονδύλια για την ανάπτυξη, για την ανάπτυξη, τότε θα αποτραπούν άλλες χώρες από το να καταπέσουν σε αυτό το χάος που έχουμε δει. Ε, δεν λέω βέβαια ότι θα σταματήσει η βία ε, στην αφετηρία της, όμως δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε κονδύλια αναπτυξιακά για ε, στρατιωτικές επιχειρήσεις ή για στρατιωτικούς λόγους εν γέννη. Αυτό μόνο. οι στρατιωτικές επιχειρήσεις χρηματοδοτούνται από κονδύλια του προπολογισμού για την άμυνα και από τα κρατη Δεν γίνεται λοιπόν να χρησιμοποιούμε άλλα κονδύλια για ε, στρατιωτικούς σκοπούς. Στην ε, χώρα μου η κυβέρνηση έχει ε, κάποιες δυσκολίες. Υπάρχουν και άλλες χώρες οι οποίες έχουν δυσκολίες στο να διαθέσουν περισσότερα κονδύλια στην άμυνα. Ορισμένες χώρες δεν έχουν λεφτά για άλλα πράγματα, πιο σημαντικά. Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφοι, πρέπει να ολοκληρώνουμε. Αυτή ήταν μία πρώτη εξέταση του σχεδίου έκθεσης. Και να σας υπενθυμίσω ότι η προθεσμία υποβολής τροπολογιών είναι η 13 Σεπτεμβρίου, 12 ώρα το μεσημέρι, αν θυμάμαι καλά. Δεύτερη εξέταση του σχεδίου έκθεσης τον Οκτώβριο. Ψηφοφορία στην Ολομέλεια Νοέμβριο, αν δεν κάνω λάθος. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Παρακαλώ να μείνετε, διότι αρχίζουμε αμέσως ε, το επόμενο θέμα της ημερησίας διάταξης. Καθίστε παρακαλώ συνάδελφοι. Μετά λοιπόν από αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων έχουμε ένα εξίσου ενδιαφέρον θέμα. Η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία. Το αποτέλεσμα της Συνόδου και οι βασικές αποφάσεις που ελήφθησαν. Θα ήθελα να καλωσορίσουμε τους ε, τρεις εκλεκτούς προσκεκλημένους μας. Τον James Απατουράη, αναπληρωτή βοηθό Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Καλώς ήλθατε. Αριστερά μου ο Διευθυντής ε, Τίμο Κώστερ, Διευθυντής της ε, Διεύθυνσης Αμυντικής Πολιτικής και Ικανοτήτων στο Τμήμα Αμυντικής Πολιτικής και Σχεδιασμού του ΝΑΤΟ. Και τέλος, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης ε, Διαχείρισης Κρίσεων και Σχεδιασμού της ΕΕΔ, Γκάμπορ Ικλόντι. Η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ εξήχθη στις 8 και 9 Ιουλίου στη Βαρσοβία, στη χώρα μου, και θα θέλαμε να ακούσουμε τους εκλεκτούς προσκεκλημένους μας για τα αποτελέσματα της ε, εκδηλώσεις, τα γεγονότα που πλαισίωσαν αυτήν την σύνοδο. Θα αναφερθούμε στην ε, δήλωση που συνυπογράφει από τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και τους ε, Προέδρους του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και από την ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπο. Δίχως καθυστέρηση λοιπόν, μια που έχουμε περιορισμένο χρόνο, θα ήθελα να δώσω το λόγο στους καλεσμένους μας. Θα αρχίσουμε με την παρουσίαση ε, από τον ε, κύριο Πατουράη. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ως ε, συνήθως Ζηλεύω όταν έρχομαι εδώ στο Κοινοβούλιο γιατί βλέπω ότι έχετε εξαιρετικά ζωντανές και ενδιαφέρουσες συζητήσεις εδώ. Όμως ε, χαίρομαι που συμμετέχω έστω και στο βαθμό στον οποίο συμμετέχω. Και οι συνάδελφοι έχουν πολλά να πούνε. Εγώ λοιπόν θα σχεδιαγραφήσω μόνο ορισμένα ζητήματα τα οποία θεωρώ σημαντικά και ενδιαφέροντα για όλους. Αρχικά την αποτροπή και άμυνα και ο Τίμο θα μιλήσει για αυτό το στοιχείο και μετά ε, το άλλο θέμα θα είναι η ε, δήλωση ε, ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αναφέρατε και εσείς. Ο συνάδελφος θα αναφερθεί επί σε αυτά τα ζητήματα. Όμως, αδρές γραμμές, θα ήθελα να σας παρουσιάσω κάποιες από τις ε, αποφάσεις στην Βαρσοβία, και γιατί ελήφθησαν. Ουσιαστικά, αρχικά έχουμε αφενός την αποτροπή στην άμυνα αφενός, και την ε, διατήρηση της ειρήνης και προβολή της ειρήνης. Για τους μάχους αυτό είναι ουσιαστικά οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, ότι δεν μπορούμε να είμαστε πλήρως ασφαλείς και προστατευμένοι στη συμμαχία μας, εφόσον δεν υπάρχει ασφάλεια και προστασία στους συμμάχους μας. Επομένω, είναι κοινό μας ε, συμφέρον ε, να βοηθήσουμε και εκείνους να διατηρήσουν την στρατητική ασφάλεια και την πολιτική τους ανεξαρτησία και αυτό αφορά και την ε, Ανατολή και τον Νότο. Θα επικεντρωθώ λοιπόν συντομία στην Ανατολή και τον Νότο και μετά θα δώσω το λόγο στους αδελφούς. Ξεκινώντας από τη Ρωσία βεβαίως γιατί πολλή από την αστάθεια στην Ευρώπη προκύπτει ουσιαστικά από τις ε, ενέργειες της Ρωσίας. Και είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι τα τελευταία 20 χρόνια το ΝΑΤΟ και όχι μόνο το ΝΑΤΟ έχουν καταβάλει πολύ σημαντικές προσπάθειες να εισαγάγουν τη Ρωσία στο ε, ευρωπαϊκό αυτό ε, και ευρωατλαντικό οικοδόμημα με σεβασμό προς τη Ρωσία αλλά και την ενθαρρύνει να είναι αξιόπιστη. Παρόλες αυτές τις προσπάθειες, ε, την συμπερίληψή της στο G7 και στο G8, στον ΠΟΕ, Παρ' όλα αυτά βλέπουμε παρόλες αυτές τις προσπάθειες ότι δεν τα καταφέραμε και εξακολουθεί να υπάρχει αστάθεια στην ε, Ευρώπη. Όπως έγινε και με την Κρυμαία, ε, τη Γεωργία, τη Μολδαβία, ε, σημαντικές επενδύσεις σε πυρηνικά προγράμματα. Πρόκειται για ένα τρομακτικό μήνυμα για τους συμμάχους και εταίρους και μια αύξηση, ένταση της στρατηγικής της παρουσίας στην Ευρώπη. Αυτό ε, οδήγησε όλους τους συμμάχους ε, στο συμπέρασμα ότι απαιτείται ανάληψη περαιτέρω ε, πρωτοβουλειών για να ενισχύσουμε ακριβώς αυτή την αποτροπή και την ασφάλεια. Τι κάναμε λοιπόν, έχουμε ενισχύσει βάσει των αποφάσεων της Βαρσοβίας. Ενισχύσαμε λοιπόν τη στήριξη για την Ουκρανία και την Κρυμαία. Αυτό θα γίνει σύντομα και για την περίπτωση της Μολδαβίας. Έχουμε εμβαθύνει την ε, συνεργασία μας με την Σοηδία και την Φιλανδία, κοινέ ασκήσεις, ανταλλαγή πληροφοριών στο στρατηγικό σχεδιασμό και ε, διαπιχειρησιακή ενίσχυση ε, σε σχέση με το παρελθόν. Σημείο εστίασης είναι και η Μαύρη Θάλασσα. Μετά τα όσα συνέβησαν στην Κρυμαία, έχουμε από πλευράς Ρωσίας ε, εντατικοποίηση της στρατηγικής της ε, παρουσίας στην Κρυμαία. Επομένω, πλέον το ΝΑΤΟ υποχρεούται να εξετάσει με μεγαλύτερη προσοχή αυτή την ε, περιοχή. Α περάσω τώρα στη Ρωσία αυτή καθ' αυτή. Είναι σαφή η προσέγγιση μα. Αφενό, διασφαλίζουμε ότι θα έχουμε την ασφάλεια για, τη, για τους συμμάχους μας, όμως θέλουμε να υπάρξει και ένα πεδίο ενίσχυσης ε, της ε, προβλεψιμότητας, της διαφάνειας, περιορισμού των ε, παρανοήσεων και ελπίζουμε κάποια στιγμή να έχουμε μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ μας. Αμφίδρομης εμπιστοσύνης. Ως συμμαχία λοιπόν έχουμε, μάλλον ξεκαθαρίσαμε αυτήν την πολιτική μας επιλογή στη Βερσοβία και εξετάζουμε το μίσο οποίο θα μπορούσαμε να έχουμε τέτοιου είδου επαγγελματικό διάλογο. Μπορούμε να, το εξετάσουμε στη συνέχεια, αν το επιθυμείτε. Στρέφουμε τώρα προ τον Νότο. Οι σύμμαχοι κατανοούν ότι το ΝΑΤΟ ω ε, οργανισμό θα πρέπει να συμβάλλει σε μεγαλύτερο βαθμό ε, ό,τι αφορά την αντιμετώπιση από τον Νότο. Στην ουσία έχουμε τρεις πυλώνες. Πρώτον πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ίδια την κρίση. Εδώ έχουμε δύο μέσα, αφενός Έχουμε το AVAX που ε, συνδράμει άμεσα ε, τον συνασπισμό. Επίσης, ήδη εκπαιδεύουμε τους Ιρακινούς αξιωματούχους. Αυτό θα γίνει, ήδη, θα γίνει πλέον και στο Ιράκ και θα ενισχυθεί για να γίνει πλέον το Ιράκ μια ασφαλής ε, περιοχή. Δεύτερος πυλώνας, να περιορίσουμε όσο γίνεται το εύρος της κρίσης. Ενισχύουμε λοιπόν τη στήριξη στην Ιορδανία, την Τινησία, εταίρους στην ε, περιοχή ε, της Μέσης Ανατολής για να μην επεκταθεί η κρίση και σε άλλες περιοχές. Και θέλουμε πάντα βεβαίως να λειτουργούμε συμπληρωματικά και να μην υποκαθιστούμε άλλες μορφές. Τρίτος πυλώνας, ε, αντιμετώπιση των επιπτώσεων, κυρίως μεταναστευτική προσφυγική κρίση. Ξέρετε ε, και την λύση που υπήρξε σε ό,τι αφορά την ε, τον περιορισμό των μεταναστευτικών ροών στο Αιγαίο και τώρα κάνουμε περαιτέρω κινήσεις ε, για τη Μεσόγειο εν γέννη. Υπήρξαν κάποιε διαβουλεύσει, τι μπορούμε να κάνουμε συμπληρωματικά ω προ την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσουμε την μεταναστευτική και προσφυγική κρίση ε, και στην υπόλοιπη Μεσόγειο. Τελευταίο μου σχόλιο, μάλλον δύο τελευταία. Πρώτον, σχέσει ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκή Ένωση υπεγράφει η κοινή δήλωση γιατί όπως αναφέρεται εκεί η ασφάλειά μας ε, η ασφάλεια και από τις δύο πλευρές ε, είναι κάτι το κοινό. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις υβριδικές απειλές με την ενίσχυση της ανθεκτικότητας, ε, επιχειρήσεις και στη θάλασσα, ικανότητες ως προς την ασφάλεια στην κυβερνοχώρο, συντονισμό σε δοκιμές και ασκήσεις και ενίσχυση της, ε, των στρατιωτικών ικανοτήτων των εταίρων μας με τον πιο έξυπνο δυνατό τρόπο για την ε, δαπάνηση των κονδύλιων μας. Το τελευταίο μου σχόλιο συνδέεται με την συζήτηση που είχατε προηγουμένω σε ό,τι αφορά τις δαπάνες, ε, τις αμυντικές δαπάνες. Είναι σαφές ότι θα πρέπει να αυξηθούν οι δαπάνες για την άμυνα στο παρελθόν που ήταν πιο σταθερά τα πράγματα και υπήρχε ασφάλεια ε, και ειρήνη, δεν χρειάζονταν ε, υψηλά κονδύλια. Πλέον όμως έχουν αλλάξει τα πράγματα. Πρέπει να επενδύσουμε λοιπόν ε, στην ασφάλεια και προστασία. Υπάρχει το ΝΑΤΟ του 2%, ο στόχος του 2% του ΑΕΠ για την άμυνα. Ο Τίμο θα σας μιλήσει ακριβώς για τα αριθμητικά στοιχεία περίπου 12 έως 16 έχουν ε, σταματήσει την περικο... τις περικοπές ε, στις αμυντικές δαπάνες. Επομένω υπάρχει μία τάση σιγά σιγά βελτίωσης αυτής της εικόνας. Και αυτό είναι θετικό. Γιατί το είπε κάποιος προηγουμένως, ότι πρόκειται για επιμερισμό του άχθους. Αυτό είναι κάτι το οποίο απασχολεί ιδιαίτερω ε, την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και όχι μόνο τον κύριο Τραμπ και ο πρόεδρος Ομπάμα έχει χρησιμοποιήσει συγκεκριμένη ορολογία για να αναφερθεί σε αυτούς που ουσιαστικά δεν ε, πληρώνουν, απλώς ε, ε, εποφελούνται του ΝΑΤΟ. Γι' αυτό και εμείς λοιπόν θέλουμε να υπάρχει μεγαλύτερη συνοχή και θα συνεχίσουμε να ασκούμε πιέσεις προς αυτό. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο, αν συμφωνείτε και εσείς Προέδρε, στον συνάδελφο. Βεβαίως, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο Τίμο Κώστερ κύριος Διευθυντής. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς ε, να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την πρόσκληση εδώ και για την ευκαιρία που μου δίνετε να απευθύνω το λόγο στην Επιτροπή σας. Νομίζω ότι είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά που έρχομαι και χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ κάθε φορά. Ο James μου διευκόλυνε πολύ το έργο μου διότι καταρχάς σας παρουσίασε την ευρύτερη εικόνα και σας εξήγησε ότι κατά βάση έχουμε δύο κύριους πυλώνες ε, που υποστήριξαν τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία. Το ένα είναι ο στόχος της ε, σταθερότητας, ε, στον οποίο αναφέρθηκε κτενός. επομένως δεν θα πω εγώ πολύ περισσότερα για τη σταθερότητα και θα μιλήσω για το δεύτερο πυλώνα, για την αποτροπή και την άμυνα. Είναι σαφές ότι το περιβάλλον ασφαλείας έχει αλλάξει και μάλιστα με διαδραματικό τρόπο τα τελευταία δύο χρόνια στην ε, σύνοδο της Ουαλίας πριν από δύο χρόνια περίπου είχαμε μια πρώτη γεύση αυτής της αλλαγής και τότε υπήρξαν ε, μία σειρά από μέτρα μέσω ε, του σχεδίου δράσης ετοιμότητας ε, όπως το αποκαλέσαμε και κάποια άμεσα μέτρα για να καθησυχάσουμε τους συμμάχους κυρίως προς Ανατολάς ότι το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να τους υπερασπιστεί εάν χρειαστεί. Είχαμε στρατεύματα και δυνατότητες διαθέσιμα και ήμασταν διατεθειμένοι να το κάνουμε. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν, μετά από τη Σύνοδο της Ουαλίας, αποφασίσαμε να, να ε, διαμορφώσουμε την ε, ε, δύναμη μάχης του ΝΑΤΟ, ενισχύθηκαν κάποια τάγματα, κάποια άλλα μειώθηκαν για να μπορούν να ανταποκριθούν σε κατεπίγουσες καταστάσεις, σε αναπτυσσόμενες κρίσεις, ουσιαστικά παντού, όχι μόνο στην, στην Ανατολική Ευρώπη, αλλά παντού. Και φυσικά αρχίσαμε να ε, κάνουμε ασκήσεις, ε, αστυνόμευση και είχαμε και πιο συχνή παρουσία στην Ανατολική Ευρώπη, κυρίως για να καθισχάσουμε τους συμμάχους μας. Έκτοτε, δυστυχώς, ε, είχαμε περαιτέρω επιδείνωση του περιβάλλοντος ασφαλείας, μια επιθετική Ρωσία η οποία παρασβιάζει σύνορα και πολλές διεθνείς συμφωνίες και η οποία δεν είναι διατεθειμένη ε, να υποχωρήσει. Η Σύνοδος λοιπόν της Βαρσοβίας ε, σε, να αυξήσει και να προσαρμόσει τις δυνατότητες αποτροπής και απάντησης του ΝΑΤΟ. Πέραν ε, αυτών των μέτρων και θα σας πω και τι προϋποθέτουν. Εξετάσαμε λίγο και τα επόμενα δύο χρόνια για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε και εκ των προτέρων ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι όχι για να μόνο για να αποστείλουμε στρατεύματα αλλά να έχουμε και κάποια σχέδια τα οποία να μπορούν να εκτελεστούν ε, πάρα αυτά. Και φυσικά ε, θέλουμε να μπορούμε να δράσουμε, όχι μόνο να έχουμε στρατιώτες οι οποίοι να μπορούν να κινηθούν γρήγορα, αλλά να έχουμε και ε, ανθρώπους οι οποίοι να μπορούν να λάβουν αποφάσεις πολύ γρήγορα εάν χρειαστεί να κινηθούμε. Τα μέτρα τα οποία συμφωνήθηκαν στην Βαρσοβία είναι αμυντικά εκφύσεως και φυσικά υποστηρίζουν ε, τις διεθνείς δεσμεύσεις ε, και τονίζουν ε, το σεβασμό των κανόνων και τη δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε αυτό, διότι πολλές συχνά μας κατηγορούν ότι είμαστε υπευθετικοί και ότι παραβιάζουμε ε, συμφωνίες οι οποίες έχουν συναυθεί στο παρελθόν. Σε καμία περίπτωση δεν ισχύει κάτι τέτοιο, σας διαβεβαιώ. Και πέραν ε, των μέτρων αυτών, όπως ε, σας είπε ο Τζέιμς ήδη, δίνουμε ακόμα μάχη για διάλογο, διαφάνεια με τη Ρωσία, μείωση των κινδύνων. Είναι λοιπόν τμήμα ε, των ε, μέτρων ε, αποτροπής και άμυνας. Είναι αναπόσπαστο τμήμα, δεν είναι κάτι το οποίο ξεχωριστό τώρα. Τι έχουμε σε αδρές γραμμές στην Σύνοδο Κορυφής στο ΝΑΤΟ. Κυρίως έχουμε σταθεί σε υποδομές και σε δυνάμεις, δυνάμεις και δυνατότητες που έχουμε ικανότητες των κρατών μελών, κάποιες ε, πολιτικές ε, και ε, κάποιες θεσμικές προσαρμογές. Καταρχάς, όσον αφορά τις δυνατότητες που έχουμε και τις ικανότητες και τις δυνάμεις μας. Οι ηγέτες αποφάσισαν για ενισχυμένη παρουσία στις χώρες της Βαλτικής και στην Πολωνία. Ο στόχος είναι να αποδείξουμε χωρίς καμία αμφιβολία ότι είμαστε αλληλέγγυοι προς τους συμμάχους, αλλά θέλουμε επίσης να ε, δώσουμε μια πραγματική απάντηση. Να μην ε, έχουμε απλώς ε, ένα μήνυμα, αλλά να μπορούμε όντως να μηνθούμε και να δράσουμε εάν προκύψει κρίση. Η πλήρης παρησία σε αυτές τις τέσσερις χώρες θα σημαίνει ότι θα υπάρχει πολυεθνικές μονάδες μάχης, οι οποίες θα παρέχονται από τέσσερις ε, χώρες ε, πλαίσιο ε, εκ περιτροπής. Θα συνεισφέρει και το ΝΑΤΟ. Οι τέσσερις χώρες οι οποίες αναλάβουν τα ενία σε κάθε μία από αυτές τις τέσσερις χώρες, τις χώρες της Βαλτικής και της Πολωνία, είναι η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ηνωμένε Πολιτείε και ο Καναδάς. Και να τονίσω εδώ ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ο Καναδάς επιστρέφει στην Ευρώπη είχαν αποχωρήσει πριν από αρκετό καιρό. Επομένως είναι πάρα πολύ ουσιαστική αυτή η κίνηση. Αυτές οι τέσσερις χώρες θα έχουν λοιπόν μια πολυεθνική μονάδα μάχης, ένα τάγμα, ε, το αποκαλούμε τάγμα συν γιατί μας επιτρέπει να υπάρχει παρουσία ανα πάσα στιγμή στις χώρες αυτές. Θα υπάρχει και ένα μικρό αρχηγείο το οποίο έχουμε ήδη συστήσει μετά από την Σύνοδο της Ουαλίας, ε, το NFRU και αυτό θα μας βοηθήσει να έχουμε μια εύρωστη παρουσία, όχι μόνο για να αποδείξουμε την παρουσία μας εκεί, αλλά και ε, θα είναι και έτοιμη για μάχη εάν υπάρξει τέτοιο θέμα. Για την ε, Νότια Ευρώπη, Ρουμανία, Βουλγαρία, την περιοχή του Ευξήνου Πόντου. Έχουμε αποφασίσει κάτι αντίστοιχο, λέγεται Taylor Forward Presence, ε, με ε, την εξής διαφορά ε, δεν έχουμε ακόμα προχωρήσει στο σχεδιασμό αυτής της παρουσίας. Ε, συζητούμε ακόμα με τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Τουρκία, τις χώρες δηλαδή ε, του Ευξήνου Πόντου, για να δούμε πώς θα σχεδιαστεί αυτή η παρουσία. Αναφερόμαστε σε θαλάσσια παρουσία στην Ευξήνο Πόντο, αλλά ίσως και ένα αρχηγείο πολυεθνικό στη Ρουμανία και ίσως και παρουσία ε, εναέρια η οποία θα πρέπει βεβαίως να αναπτυχθεί περαιτέρω. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τη στρατιωτική μας παρουσία και τις δυνάμεις μας. Θα ήθελα να τονίσω ότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ε, συμφώνησαν ότι το ΝΑΤΟ έχει όλες τις ικανότητες που είναι απαραίτητες για να ε, σχεδιάσει όλες αυτές τις αποστολές της συμμαχίας. Πέραν λοιπόν ε, της οικονομικής δέσμευσης που θα αναφέρω λίγο αργότερα, είναι μια πολύ σημαντική δέσμευση η οποία πηγαίνει πολύ πέρα των δυνάμεων που έχουμε ε, αυτή τη στιγμή. Έχουμε όλες τις ικανότητες, ε, όλες τις ε, αποστολές που αποτελούν δέσμευση για τους ηγέτες και είναι διαθέσιμα τα στρατεύματα. Τώρα, όσον αφορά την παρουσία που έχουμε σε διάφορα χώρες της συμμαχίας. Καταρχάς, ο Τζέιμς αναφέρθηκε σε αυτό. Υπάρχει ένα πλαίσιο για την απάντηση του ΝΑΤΟ στις ε, διάφορες απειλές ε, και προκλήσεις που υπάρχουν ε, από τον Νότο, πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε και τι μπορούμε να κάνουμε για τα διάφορα θέματα στον Νότο. Υπάρχει μια στρατηγική για ε, ανταρτοπόλεμο, υβριδικό ανταρτοπόλεμο σε κάθε χώρα. Ε, όπως είπε και ο Τζέιμς, αυτό αφορά συνεργασία μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά οι επικεφαλείς της συμμαχίας ε, ε, συμφώνησαν για τη λεγόμενη δέσμευση για την κυβερνοάμυνα και θέλουν να ενισχύσουν τα δίκτυα της κυβερνοάμυνας ε, της κάθε χώρας ως προτεραιότητα. Επίσης, εθνική αντοχή για κάθε χώρα που περιλαμβάνει και την κυβερνοάμυνα. Και επίσης, ένα πολύ σημαντικό θεσμικό ε, ζήτημα, οι επικεφαλείς ε, των κρατών και κυβερνήσεων συμφώνησαν ότι θα επανεξετάσουμε ε, την ε, δομή της ηγεσίας του ΝΑΤΟ. Ξέρετε ότι ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ΝΑΤΟ είναι ότι υπάρχει ε, μία μόνιμη ηγεσία με αρχηγία σε διάφορα σημεία, δυνατότητες και ικανότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την αντίστοιχη ηγεσία και έχει εξελιχθεί αυτή η ηγεσία. Η τελευταία εξέλιξη ήταν το 2010, αλλά έκτοτε έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Το 2010 έγινε μια μεταρρύθμιση με την πολύ σημαντική πρόθεση να μειωθεί το κόστος και το μέγεθος και η μορφή ε, της ηγεσία. Αυτή τη στιγμή βέβαια είμαστε στην αρχή της νέας μεταρρύθμισης, αλλά να σας πω ότι η πρόθεσή μας είναι να επαναφέρουμε μια σειρά από ικανότητες ε, σε, αυτή τη δομή ηγεσία και φυσικά αυτό σημαίνει ότι το μέγεθος και η σύνθεση κατά πάσα πιθανότητα θα αυξηθούν. Ε, την επόμενη διετία, ώστε να είμαστε σε θέση να κάνουμε κάτι το οποίο φανταστείζόμασταν ότι δεν θα χρειαζόμασταν να ξανακάνουμε ποτέ, να αντιμετωπίσουμε πιθανό πόλεμο στην Ευρώπη. Είναι πολύ σημαντική πρόβλεψη αυτή για τις ε, δομές της ηγεσία του ΝΑΤΟ. Από πλευρά μου τώρα να πω και κάτι τελευταίο για την ε, επενδύσεις ε, στην άμυνα κάθε σύμμαχος θα πρέπει να δαπανά 2% ε, του εθνικού του προϋπολογισμού στην άμυνα. Αυτή είναι μια δέσμευση η οποία αναλήφθη στην ε, Σύνοδο Κορυφής της Ουαλίας, ε, στην Σύνοδο της Βαρσοβίας επιβεβαιώθηκε αυτή η δέσμευση και επίσης έγινε και μια εξέταση της κατάστασης και με κάποια ικανοποίηση είδαμε ότι υπάρχει αύξηση στις αμυντικές δαπάνες στους 16 από τις 28 χώρες. Αυτή τη στιγμή νομίζω 6 χώρες ε, ε, που είναι ε, πάνω από το 2% και το πιο σημαντικό είναι ότι οι περισσότεροι σύμμαχοι κατάφεραν να αυξήσουν την παραγωγή. Δηλαδή δεν είναι μόνο ε, τα όσα διαθέτεις στον προπολογισμό για την άμυνα, αλλά και σε τα δαπανάς. Θα τα δαπανάς σε πράγματα τα οποία απαιτεί το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο ή αφορά μόνο ικανότητες του ΝΑΤΟ, αλλά το θέμα είναι και αν θα διατίθενται αν τα χρειαζόμαστε. Γιατί τι να το κάνεις να έχεις στρατεύματα και εξοπλισμούς εάν δεν τα διαθέτει ε, στις αποστολές του ΝΑΤΟ. Θεωρώ ότι αυτή είναι μια ταπεινή ιστορία επιτυχίας, ε, σαφώς μπορεί να γίνουν πολύ περισσότερα. Πρέπει να συνεχίσουμε τις πιέσεις και θα έλεγα όχι μόνο από πλευράς ΝΑΤΟ αλλά και από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στο 80% αναφερόμαστε στο, ε, ίδιο, στις ίδιες δαπάνες και το ίδιο εκλογικό σώμα που πρέπει να υποστηρίξει τους ηγέτες μας. Θα σταματήσω εδώ και θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, συγγνώμη που πρόφερα το όνομά σας λάθος, κύριε Κλώδη. Μάλλον φταίει το ότι είμαι γιατί ταξίδευα πολύ νωρίς. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Είναι πάντα μεγάλη χαρά να έρχομαι στην Επιτροπή σας. Οι συνάδελφοί μου μίλησαν και άφησαν ελάχιστα για μένα. Και πραγματικά υπάρχουν ελάχιστα που μπορώ να πω χωρίς να επαναλάβω αυτά που είπατε. Θα προσπαθήσω όμως να επικεντρωθώ σε δύο πράγματα, αλλά ας αρχίσω από αυτό που συνηθίζεται, δηλαδή ότι όποτε γίνεται μία σύνοδος του ΝΑΤΟ, πάντα καλείται η, η υπατή εκπρόσωπος ε, Φεντερίκα Μογκερίνη. Και είναι πάντα παρούσα. Είναι λοιπόν σημαντικό να διατηρηθεί αυτή η παράδοση και στο μέλλον, έτσι ώστε οι σύνοδοι του ΝΑΤΟ να περιλαμβάνουν και ένα διάλογο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, να υπάρχει διάλογος ανάμεσα στους αρχηγούς και των δύο είναι, οργανισμών. Είναι επίσης σημαντικό για να στείλουμε και το μήνυμα της καλής συνεργασίας. Επίσης, η ατζέντα μας είναι παρόμοια. Όλοι μιλάμε για τις δαπάνες της άμυνας, για την αύξηση ικανοτήτων. Αυτό έγινε και στην ε, δικοινοβουλευτική συνάντηση στην Πρατισλάβα, όπου η Φεντερίκα Μοκερίνη αναφέρθηκε στα θέματα που ε, άπτονται της ε, άμυνας μετά από τον έλεγχο της ε, υλοποίησης του θεματολογίου για την άμυνα. Είναι λοιπόν τα ίδια θέματα που απασχολούν και τους δύο οργανισμούς. Καταρχάς η κοινή δήλωση, εκτός του ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό πολιτικά και για τους δύο οργανισμούς. Ε, στέλνουμε δηλαδή ένα μήνυμα ότι ενώνουμε τις δυνάμεις μας και αντιμετωπίζουμε ενωμένοι ε, τα προβλήματα δεν είναι μόνο όμως αυτό, δεν είναι μόνο η κοινή δήλωση την οποία έχουν συμφωνήσει οι επικεφαλείς των δύο οργανισμών, ο πρόεδρος Γιούγκερ, ο πρόεδρος Τούσκ και ο κύριος Τόλτεμπερκ από το ΝΑΤΟ. Ο μηχανισμός υλοποίησης είναι ε, κάτι που παρουσιάστηκε πλέον, κάτι το οποίο θα ασκήσει πίεση και σε εμάς για να Υποβάλλουμε αυτήν την έκθεση προόδου το Δεκέμβριο, μια έκθεση προόδου για θέματα ε, τα οποία ακούσατε μόλις, τι έχουμε δηλαδή επιτύχει. Και επίσης ασκεί πολιτική πίεση στους ε, δύο οργανισμούς για να υποβάλουν τακτικές εκθέσεις προόδου. Τι έχει επιτευχθεί. Στους τομείς που ακούσατε από τους συναδέλφους όπως ε, ανέφερε και ο James, υβριδικές απειλές, κάτι το οποίο ακούσατε. Νομίζω πως θα έχουμε τη δυνατότητα μέχρι το Δεκέμβριο να δείξουμε ουσιαστικά αποτελέσματα στον, ΕΘΕ, στον τομέα αυτό. Αυτό που ονομάζει το NATO Playbook, επιχειρησιακό πρωτόκολλο, είναι σημαντικό να δούμε το πλαίσιο, να δούμε ε, τα σημεία επαφής των δύο οργανισμών μέσω των οποίων θα επικοινωνούν για τέσσερις βασικούς ε, τομείς. Καταρχάς η επαγρύπνηση. Όπως θα γνωρίζετε, έχει επίσημα δοθεί η έναρξη αυτών των υβριδικών μορφών, των υβριδικών κιτάρων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημοσιεύσει 24 έγγραφα μέχρι τώρα. Μετά, πρόληψη κρίσεων και απάντηση σε περιπτώσεις δηλαδή κρίσεων δεν θα μπορούμε μόνο να εντοπίζουμε αυτές τις κρίσεις αλλά να απαντούμε και καταλήλως. Αυτό είναι το καλύτερο που μπορούμε να δώσουμε στα κράτη-μέλη, να δώσουμε δηλαδή μια καλή συνεργασία ανάμεσα ε, στους οργανισμούς. Μετά, κυβερνοάμυνα. Είναι πολύ σημαντικό τομέας και κοινωνικά και οικονομικά. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό ε, όχι μόνο για τους γείτονές μας, αλλά και για εμάς τους ίδιους να υπάρχει εναρμόνιση των υπηρεσιών πληροφοριών. Τώρα, στη θάλασσα είναι πολύ σημαντικό, όπως είδαμε και τους τελευταίους μήνες, να υπάρχει καλή συνεργασία. Είδαμε την, ε, το παράδειγμα του Αιγαίου, τον συντονισμό των δραστηριοτήτων του ΝΑΤΟ και της Frontex. Το σημαντικό είναι εδώ ότι καταφέραμε να σπάσουμε ορισμένους φραγμούς ε, επικοινωνιακής φύσης. Προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε και το καταφέραμε τα προβλήματα στην ανταλλαγή πληροφοριών αυτή η κοινή ε, άσκηση των δύο υπηρεσιών απέδειξε ότι υπάρχει τρόπος για να το καταφέρουμε αυτό. Επίσης, θεωρώ ότι ακόμα σημαντικότερη θα γίνει η δραστηριότητα στη Μεσόγειο μέσω μιας εντολής που θα συμπεριλαμβάνει και ε, μετακπαίδευση της ακτοφυλακής για ε, θέματα διακίνησης όπλων. Για το ΝΑΤΟ είναι μια πολύ καλή συνεργασία και για την ανταλλαγή πληροφοριών και για τις αναγνωριστικές ε, δραστηριότητες και για όλο τον ε, συντονισμό των επιχειρήσεων. και πιστεύω πως ε, βασισμένη σε αυτό θα σχεδιαστεί και η μελλοντική μας στρατηγική. Και στόχος μας θα είναι να φροντίσουμε να διαχειριστούμε τους πόρους κατάλληλα χωρίς να αφήσουμε ε, κενά τα οποία θα μας κοστίσουν στο μέλλον. Έπειτα, οι κυβερνοπηλές Πιστεύω δεν χρειάζεται να σας αναφέρω πόσο σημαντικό είναι να συνεργάζονται οι δύο οργανισμοί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Όπως γνωρίζετε, ε, ψηφίστηκε η σχετική οδηγία, έχει τεθεί σε ισχύ και είναι ένα βασικό μέσο για να αυξηθεί η ανθεκτικότητα στα κρατημέλη. Καλύτερη προστασία δηλαδή στον κυβερνοχώρο και αυτό είναι καλό και για το ΝΑΤΟ. Και πιστεύω εδώ η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν σημαντικότατη. Φυσικά υπάρχουν και άλλα που μπορούν να γίνουν. Τυποποίηση, για παράδειγμα, των ε, προϋποθέσεων ανάπτυξης ε, στρατιωτικών μονάδων. Τώρα, άμυνα, αμυντικές ικανότητες. Θα μας απασχολήσει πολύ στο μέλλον ο αμυντικός σχεδιασμός. και θα γίνεται λόγο στα πλαίσια του ε, EUGS η ανάπτυξη στρατιωτικών ικανοτήτων τις οποίες θα χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και για τις δικές της αποστολές και για τις αποστολές που θα γίνουν σε συνεργασία με το ΝΑΤΟ. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να ε, προβλεφθούν όλες οι ανάγκες. Ένας πολύ σημαντικός τομέας ε, αυτού είναι και το λιμενικό θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο και στο μεταναστευτικό θέμα και στην φύλαξη των συνόρων. Η αύξηση δηλαδή των ικανοτήτων του λιμενικού. Αμυντικές ικανότητες τώρα, αμυντική βιομηχανία, έρευνα, το Ευρωπαϊκό Σχέδιο ε, Δράσης για την Άμυνα, EDAP, θα μας απασχολήσει πολύ. Οι διάφορες ε, κοινέ ασκήσεις. Προσπαθούμε να ε, συγχρονιστούμε στις ασκήσεις μας, να κάνουμε κοινέ ασκήσεις ή δυνατόν, πολιτικές ασκήσεις, ιδιαίτερα ε, ασκήσεις που αφορούν υβριδικές ασκήσεις. Προσπαθούμε λοιπόν να τις διεξάγουμε σε ένα κοινό περιβάλλον Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ και όχι ε, ο καθένας ξεχωριστά. Διότι όλα πρέπει να είναι αποτέλεσμα συνεργασίας από την ε, πρόληψη, την αποτροπή, την αντιμετώπιση. Τέλος, ε, το θέμα των εταίρων είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους εταίρους μας. Με πολλούς τρόπους με την κοινή μας παρουσία, η Ορδανία, η Ιράκ, αλλά και στην Ανατολή, στα Ανατολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Γεωργία, τη Μολδαβία. Είναι πολύ σημαντικό να ε, συντονίσουμε τις ε, προσπάθειές μας. Επίσης, ε, γι' αυτό θα μας βοηθήσει και η αναθεώρηση της ε, πολιτικής γειτονίας. Κάτι το οποίο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και θέματα ασφαλείας και πρέπει να περιλαμβάνει και τη δυνατότητα ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της ασφάλειας. Αυτό θα είναι πολύ σημαντικό στο μέλλον. Πιστεύω λοιπόν πως υπάρχει μια πληθώρα τόμεων που μπορούμε να συνεργαστούμε. Υπάρχουν τα μέσα, αυτή η κοινή δήλωση η οποία θα διασφαλίσει αποτελέσματα μέσα σε ένα χρονικό πλαίσιο το οποίο θα συμφωνηθεί και υπάρχει και η πολιτική εποπτεία η οποία θα πρέπει να ε, συζητηθεί από εμά. Θα σταματήσω όμως εδώ και θα σας δώσω το λόγο κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Διευθυντά. Ο κύριος Γκάλερ, πρώτος ε, ομιλητής εκ των Ευρωβουλευτών. Ευχαριστώ πολύ. Ξενόμετος της ομάδας ε, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ευχαριστώ και για τις τρεις παρουσιάσεις. Εν γέννη, θεωρώ ότι είναι ικανοποιητικό το αποτέλεσμα της Συνόδου Κορυφή του ΝΑΤΟ. Έχουν αποσταλεί σαφή μηνύματα. Και από ό,τι φαίνεται υπάρχει και η πολιτική βούληση για να υλοποιηθούν τα απαραίτητα. Κοιτάζοντας τον Ευρωπαϊκό Χάρτη και τον τελευταίο αιώνα πιο συγκεκριμένα, η εμπειρία δείχνει ότι οι σταθερές δημοκρατίες τείνουν να μην είναι επιθετικές ή προσβλητικές προς ε, τους ε, γείτονες ούτε μεμονωμένα, ούτε συλλογικά, ούτε και ομόφωνα, όπως είναι ο τρόπος που αποφασίζει το ΝΑΤΟ. Έτσι, ακόμα και στο παρελθόν που υπήρχε η Σοβιετική Ένωση, μπορούσαν να είναι σίγουροι ότι δεν υπήρχε καμία τέτοια απειλή από πλευρά μα για στρατιωτική ανάληψη ε, στρατιωτική ε, παρέμβαση. Υπήρχε μόνο η πρόκληση ε, ενό δημοκρατικού παραδείγματο. Μόνο αυτό του απειλούσε. Σήμερα λοιπόν έχουμε την πρόκληση διαμόρφωση τη πολιτική βούληση για να περασπιστούμε όχι μόνο τα ιδανικά μα, αλλά και την επικράτειά μα. Υπήρχε υπήρχαν αυτές οι περικοπές ε, στις αμυντικές δαπάνες στις τελευταίες δύο δεκαετίες. Επομένω, αυτή η βούληση αντιμετώπισης της πραγματικότητας ε, βλέπουμε ότι είναι δύσκολες ε, για την κοινωνία μας. Ορισμένοι λοιπόν προσπαθούν να υποτιμήσουν ή και να αγνοήσουν τις προκλήσεις. Όμως νομίζω ότι το ΝΑΤΟ έδωσε κατάλληλη απάντηση. Σε ό,τι αφορά αυτό τον όρο συμπληρωματικέ ενέργειε που έχει αναφερθεί και στην κοινή δήλωση. Έχω ένα ερώτημα. Πώς έχουν οι συζητήσεις σε ό,τι αφορά τη στήριξη, οικονομική στήριξη άλλων τέτοιων ενεργειών από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Έχω πει και σε άλλες περιστάσεις ότι αν αποφασίσουμε σε επίπεδο ΝΑΤΟ να έχουμε επιπλέον στρατιωτικές δυνάμεις, Λετωνία, ε, Λιθουανία, Πολωνία έχει γίνει αυτό, αλλά και πρακτικά εγκαταστάσει, διαμονή. Γιατί αυτό να αφορά μόνο τις ε, εν λόγω χώρες είναι κάτι το οποίο αφορά όλους μας, το κοινό μα συμφέρον. Επομένω θα μπορούσε να υπάρξει κοινοτική χρηματοδότηση σε ό,τι αφορά την ε, οικοδόμηση αυτών των εγκαταστάσεων ή ακόμα και ηρωνικά ε, να πούμε ότι μπορούμε να αναπαλαιώσουμε παλιά σοβιετικά στρατόπεδα και ούτω καθεξής. Πρόκειται για υποδομές που όχι σκόπουμε βέβαια, αλλά de facto μας επηρεάζει όλους. Αυτό αφορά και τις ε, διόδους μεταφορών. Θέλουμε να έχουμε έναν, ε, μια ευρωπαϊκή τέτοια οδό μέσω Πολωνίας και Λιθουανίας. Υπάρχει ένας τέτοιος σχεδιασμός, αλλά θα μπορούσε να επιταχυνθεί αυτός ο σχεδιασμός και μετά ως επιπλέον όφελος σε περίπτωση ανάγκης θα μπορούσε ακριβώς, ε, ε, αν χρειαστεί και πάλι επισημένο, να ε, χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά στρατιωτικών δυνάμεων. Μπορούμε λοιπόν να σκεφτούμε λίγο δημιουργικά για να δούμε τι μπορούμε ακριβώς να κάνουμε. Έχετε εσείς τέτοιου είδους σκέψεις. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριο Σκάν. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ και τους ε, τρεις ομιλητές. Και να πω ότι χαιρετίζουμε αυτή τη συνεργασία και που βλέπουμε τώρα ε, μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαίρομαι που έχει πλέον κληθεί και το ε, Μαυροβούνιο για να γίνει το 21ο μέλος της Συμμαχίας. Υπάρχουν σχέδια για τη συμπερίληψη άλλων βαλκανικών χωρών, για παράδειγμα η Βοσνία. Τώρα για την νότια γειτονία. Μιλήσατε για μια σειρά ενεργειών που έχετε αναλάβει που και πάλι είναι θετικές. Το ερώτημα που έχω είναι ποιες θεωρείτε ότι είναι οι δυνατότητες που έχει εδώ ο ISIS. Βλέπουμε ότι έχουν υποχρεωθεί να αναδιπλωθούν σε ό,τι αφορά τις εκτάσεις που κατήχαν στο Ιράν και στη Συρία. Πού βρίσκομαστε λοιπόν και υπάρχει αυτή η απειλή του κατακαιρματισμού του ISIS και πώς αυτό μάλλον απειλεί εμάς ε, στη συνέχεια. Μετά, δεν ξέρω αν θα μπορούσατε να σταθείτε εν συντομία και στην κατάσταση στο Αφγανιστάν. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια επιδείνωση και εκεί. Υπάρχει κάτι καινούργιο που μπορούμε να κάνουμε, γιατί συμμετέχουμε εκεί τόσα χρόνια, αλλά βλέπουμε ότι δεν επιτυχάνεται η επιθυμητή πρόοδος. Άλλα τέτοια διδάγματα είδαμε στο Ιράκ, σε ό,τι αφορά την κατάρτιση και εκπαίδευση των ε, αξιωματούχων και θεωρητικών δυνάμων. Είδαμε όμως τι έγινε εκ των υστέρων όταν υπήρξε πίεση από τον Άισις. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βανόρντεν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και πάντα χαίρομαι ιδιαίτερα όταν βλέπω εκπροσώπους ε, της ε, Συμμαχίας του ΝΑΤΟ εδώ στην ε, Επιτροπή μας. Πάντα λυπάμαι που το ΝΑΤΟ αναγκάζεται να παίξει το παιχνίδι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιλαμβάνομαι γιατί, γιατί έχετε εκπροσώπους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά και τον εκπρόσωπό μας ε, στο ε, Βορειοατλαντικό Συμβούλιο και ξέρουμε πώς ε, γίνεται η επικοινωνία από σύνοδο σε σύνοδο. Θα υπάρχουν τουλάχιστον τρεις χώρες οι οποίες θα επιμένουν να αναφέρεται ο ρόλος Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλα τα συναφή. Κρίμα, διότι όσο περισσότερο ενθαρρύνεται αυτό το παιχνιδάκι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο περισσότερο χάνεται ενέργεια, πνευματική ενέργεια και όλη αυτή η διαδικασία συγχρονισμού, συντονισμού και όλα αυτά τα πράγματα είναι σπατάλη προσπάθειας. Στην πραγματικότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κανέναν απαραίτητο ρόλο όσον αφορά την άμυνα. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει κάποια χρήσιμα πράγματα από πολιτική σκοπιάς. Αυτό να το αναγνωρίσω αλλά φυσικά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συμμετέχει σε αυτό το παιχνίδι, έχει φιλοδοξίες άμυνας και λυπάμαι που γίνεται οτιδήποτε ε, που ενθαρρύνει τα πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί αυτά είναι εις βάρος του ΝΑΤΟ. Γιατί ούτως ή άλλως αναφερόμαστε στις ίδιες χώρες και είναι γελίο να πρέπει να συγχρονίζουμε τις προσπάθειες ε, των ίδιων χωρών τελικά. Να αναφερθώ σε κάποια συγκεκριμένα ζητήματα. Καταρχάς, η επιχείρηση για τους πρόσφυγες στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο. Νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα προβληματικά τα πράγματα εκεί. Ένα κοινικό θα μπορούσε να πει «Ε, γιατί να μην στήσουμε φέρει από τη Βόρεια Αφρική να εκδίδουμε εισιτήρια και να περνάνε απέναντι. Γιατί περνάμε ε, από όλη αυτή την φάρσα να περιμένουν να πνίγονται στη Μεσόγειο και μετά να τους σώζουμε. Η ερώτησή μου είναι ποια είναι η σωστή χρήση των στρατιωτικών και ναυτικών ε, δυνάμεων του ΝΑΤΟ σε αυτές τις επιχειρήσεις. Θεωρούμε ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Κάτι άλλο το οποίο θα ήθελα να τονίσω, το οποίο ανέφερε ακροθυγός ο Τίμο, είναι η Τουρκία. Είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα. Πολλοί από εμά εκτιμούν την Τουρκία ως έναν πολύ ισχυρό ε, μέλος της συμμαχίας του ΝΑΤΟ και από γεωγραφική σκοπιά είναι σε στρατηγική θέση, είναι πάρα πολύ σημαντική η δουλειά που κάνει η Τουρκία. Και θα ήθελα να ξέρω, δεδομένου ότι υπάρχουν δυσκολίες αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν σχέσεις με τον Πούτιν και τη Ρωσία, υπάρχει το θέμα της συνοχής και της ε, συνέπειας της συμμαχίας ε, στις μεγάλες επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ που ασχολείται με τα προβλήματα στη Συρία, επί παραδείγματι. Και σε ποιο βαθμό ε, τα οδηγούμε όλα αυτά προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα ήθελα όμως να, πω λίγα περισσότερα, να ακούσω λίγο περισσότερα για την Τουρκία ως σύμμαχό μας. Ευχαριστώ η κυρία Λουίζινγκ. Σας ευχαριστώ πολύ. να αναφοράσετε τα ακουστικά σας παρακαλώ. Έχω τρεις ερωτήσεις. Καταρχάς, σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για τις παρουσιάσεις σας. Στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ αναφέρθηκε η χρησιμοποίηση του ΕΒΕΞ για την, για το, στον πόλεμο κατά του Ισλαμικού κράτους. Δεν ακούσαμε όμως κάτι μετά από αυτό. υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες, τι έχει αποφασιστεί για το ρόλο της ε, Τουρκίας, για το τι κάνει η Τουρκία με, με τους ε, Κούρδους. Τι γίνεται λοιπόν με το ΑΒΑΞ. Μετά, Αφγανιστάν. Υπάρχει μια συγκεκριμένη ημερομηνία για το τέλος ε, της αποστολής, διότι αναβάλλεται. Οι αναβολές είναι συνεχόμενες, δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο τέλος και εάν κατάλαβα καλά δεν υπάρχει λοιπόν κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία αποχώρησης των στρατευμάτων. Τι συμβαίνει λοιπόν, ποιο είναι το πλάνο. Μετά αναφέρθηκε από κάποιον συνάδελφο η Ανατολική Ευρώπη και η επανέναρξη του διαλόγου με τη Ρωσία έτσι ώστε να δημιουργηθεί εκ νέου εμπιστοσύνη. Αυτό λοιπόν αποφασίστηκε στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Εγώ δεν μπορώ να βρω ακριβώς ε, πώς θα οικοδομηθεί ξανά εμπιστοσύνη. Μπορείτε ίσως να μας ενημερώσετε για το τι μελγενέστε από αυτού. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τις ε, παρουσιάσεις σας. Είναι πολύ σημαντική, πιστεύω, αυτή η σύνοδος ε, στην Βαρσοβία. Η σύνοδος γίνεται κάθε δύο χρόνια και πιστεύω ότι ήταν και πολιτικά σημαντική. διότι οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν και πολιτικού χαρακτήρα, όχι μόνο στρατιωτικού χαρακτήρα, ιδιαίτερα για ε, αυτά που συμβαίνουν στα ανατολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά τα κράτη-μέλη είναι διαφορετικά επηρεασμένα από τις εξελίξεις, όμως υπάρχει η ετοιμότητα, η διάθεση για συνεργασία. Πολιτικά ε, τουλάχιστον αυτό απεδείχθη από την ε, Σύνοδο. Και πιστεύω πως η Πολωνία ως ε, οικοδεσπότη ήταν, ήταν πάρα πολύ καλά προετοιμασμένη. Δεν μπορώ να πω όμως πως είμαι σίγουρος για το αν είναι αναλογική μία στρατιωτική απάντηση, μία στρατιωτική παρέμβαση. Και δεν είμαι σίγουρος κιόλας εάν θα είναι στρατιωτικά επαρκής αυτή η λύση αυτά τα στρατεύματα για τα οποία έγινε λόγος δεν είναι τα τυπικά στρατεύματα. Οι δομές τους είναι διαφορετικές. Θα αποτελούνται από στρατιώτες των Ηνωμένων Πολιτειών αυτές οι μονάδες. Από ποιους θα αποτελούνται. Επίσης θα χρησιμοποιείτε όλο το δυναμικό αυτών των ε, μονάδων ή κάποιο ποσοστό από αυτό 40-50%. Τι, τι θα γίνει με τη σύσταση λοιπόν, πώς θα είναι δομημένες αυτές οι μονάδες, θα μπορούν να δράσουν άμεσα ή θα χρειαστούν περισσότεροι μεταφραστές, περισσότεροι διερμηνείς για δεδομένη στη συμμετοχή πολλών χωρών. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο θέμα. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω. Ε, κάτι που με ανησυχεί. Αν κοιτάξουμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο ΝΑΤΟ και τι κάνει η Ρωσία, θα δούμε ότι το ΝΑΤΟ προετοιμάζεται για περισσότερες ασκήσεις, οι οποίες θα είναι ευρύτερες. Στην Πολωνία, μάλιστα, θα ε, κινητοποιηθούν 30.000 στρατιώτες στα πλαίσια αυτών των ασκήσεων. Η Ρωσία από την άλλη έχει ε, μία προσέγγιση δύο ε, κατευθύνσεων και ασκήσεις αλλά και άμεση αντίδραση χωρίς προειδοποίηση, χωρίς ανακοίνωση με μετακίνηση περίπου 100.000 στρατιωτών μέσα σε μια νύχτα. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε τι δυνατότητες έχουμε σε περίπτωση που εμφανιστεί μία κρίση. Και τρίτον, κοίταξα τα έγγραφα τα οποία ψηφίστηκαν στη Βαρσοβία και μπορώ να πω ότι τα διάβασα προσεκτικά και με ανησυχεί το ε, θέμα των υποδομών, NSAP. Εάν για παράδειγμα θέλουμε να κινητοποιήσουμε 40.000 στρατιώτες άμεσα, δεν θα είναι μόνοι τους, θα έχουν οπλισμό, θα έχουν πολλά παρελκόμενα. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι θα γίνει με τις επενδύσεις στα υποδομών στα ανατολικά. Δεν εννοώ μόνο τα αεροδρόμια. Μιλώ για γενικότερες υποδομές, οι οποίες δεν είναι επαρκώς χρηματοδοτημένες. Ε, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους κύριους ομιλητές ε, για τις παρεμβάσεις τους. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για την καθυστέρηση. Αλλά υπήρχαν ανελημμένες υποχρεώσει. Δεν άκουσα λοιπόν την πρώτη ομιλία και ζητώ συγγνώμη. Έχω ένα πολύ σύντομο και απλό ερώτημα. για τα όσα ανέφερε ο κ. Κώστερ. Στο τέλος ουσιαστικά της ε, παρέμβασής του. Από τις σημειώσεις μου βλέπω ότι αναφέρεστε στο γεγονός ότι το ΝΑΤΟ έχει περιορίσει τα στοιχεία, τα οικονομικά στοιχεία, κατά, σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον, ε, σε ό,τι αφορά τα κονδύλια που διατίθενται συνήθως. Και μετά είπατε ότι κάτι έπρεπε να κάνουμε που μάλλον αναγκαστήκαμε να κάνουμε κάτι το οποίο θεωρούσαμε ότι δεν θα χρειαστεί πλέον να το κάνουμε, να πολεμήσουμε στην Ευρώπη. Και πραγματικά εξεπλάγει από αυτή τη δήλωση, από αυτή τη διατύπωση. Να διεξάγουμε πόλεμο στην Ευρώπη, είπατε. Αυτό δεν αφορά και τους άλλους από την άλλη πλευρά που διατείνονται ότι η αποστολή τους πάντα ήταν και πάντα θα είναι να κάνουν ακριβώ αυτό. Δηλαδή να διεξάγουν ένα πόλεμο στην Ευρώπη. Μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο αυτή σας ε, την πρόταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν έχει ζητήσει κανεί άλλο το λόγο. Να κάνω λοιπόν και εγώ τα δικά μου ερωτήματα, αν επιτρέπετε. Γιατί και εγώ μία απλή ευρωβουλευτή είμαι. Ο κύριος Βανόρντεν έχει ήδη θέσει το πρώτο ερώτημα που ήθελα να κάνω κι εγώ. Ε, ήθελα κι εγώ να σταθώ στο ζήτημα της Τουρκίας. Την κατάσταση εκεί. Δεύτερον, υπήρξαν σημαντικές ανακοινώσεις από διμερείς συνεδριάσεις με τη Γεωργία και την Ουκρανία στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής, ε, με ελαφρώς διαφορετική διατύπωση από ό,τι παρατήρησα. Θα ήθελα λοιπόν και τη δική σας γνώμη σε ό,τι αφορά τη συνέχεια που θα δοθεί σε αυτό. γιατί εστιάζουμε την προσοχή μας σε, τόσο διαφορετικ... σε τόσους διαφορετικούς τομείς και ανεξάρτητα από τις προσπάθειές μας βλέπουμε ότι η Ουκρανία πόρο απέχει και από τη σταθερότητα ακόμα. Γιατί υπήρξαν ε, απίστευτα γεγονότα, αποτρόπαια εγκλήματα, ε, βομβαρδισμοί, ε, μεγάλος αριθμός θυμάτων, αμάχων από, τους, από τις απο, αποκαλούμενες αποσχιστικές ε, δυνάμεις, αλλά σε μια δύσκολη και αμφισβητήσιμη κατάσταση, είναι και περισσότερο μάλιστα, σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κρυμαία. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν ε, για να δοθεί συνέχεια σε αυτά τα ανακοινοθέντα. Να αρχίσουμε από εσάς ε, τις απαντήσεις. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για όλα τα εξαιρετικά ενδιαφέροντα αυτά ερωτήματα και χαίρομαι που έχω τη δυνατότητα να απαντήσω σε ορισμένα από αυτά. Βεβαίω, οι συνάδελφοι είναι και πλέον οι δήμονε σε αρκετά από αυτά τα θέματα. Δεν θα αναφερθώ στον ε, προπολογισμό το κοινοτικό, θα μιλήσω όμω ε, συντομία για τα Βαλκάνια. Υπάρχουν δύο ακόμα βαλκανικέ χώρε που φιλοδοξούν να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. για να είμαστε ειλικρινεί και στι δύο αυτέ περιπτώσει υπάρχουν σημαντικέ προκλήσει πολιτική φύσεω, ό,τι αφορά το εσωτερικό πολιτικό του σκηνικό. Το ΝΑΤΟ έχει θέσει πολύ συγκεκριμένα κριτήρια ε, για να μετρήσουμε την πρόοδό τους ε, και τους έχουμε ενθαρρύνει, αλλά από εκεί πέρα δεν μπορούμε να ε, επηρεάσουμε και πολλά τα πράγματα. Για τον ISIS ε, έχετε θέσει ένα εξαιρετικά σύνθετο ζήτημα για τις ε, ικανότητες του ISIS και τι θα γίνει στη συνέχεια. Είναι μια μακροσκελής απάντηση αυτή. Υπάρχουν και μάλιστα πολλές διαφορετικές απαντήσεις. Και το αναλύουμε συνεχώς. Να σας πω δύο πράγματα. Πρώτον, υπάρχει πρόοδος στο Ιράκ στη Λιβύη, όχι πέρα από εμάς, στην αντιμετώπιση του ISIS ως μιας παραδοσιακής στρατιωτικής δύναμης που κατέχει επικράτεια, εδάφη. Υπάρχει πρόοδος ότι αφορά ε, των περιορισμών της χρηματοδότησης του ISIS, αλλά και σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του προσελητισμού ε, και της προσέλκυσης μελών. Τη στρατολόγηση μελών. Υπάρχει λοιπόν σημαντική επιτυχία και πρόοδο εδώ. Από την άλλη βέβαια ισχύει ότι ο ISIS έχει πλέον ε, διαμορφώσει δεσμούς με άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις, Al-Shabaab, Boko Haram, 7 με 12 άλλες τρομοκρατικές, τρομοκρατικές οργανώσεις μάλιστα θα έλεγα. Ακόμα και αν στρατιωτικά λοιπόν ιτώνται, βλέπουμε ότι είναι ένα μακροπρόθεσμο πρόβλημα το οποίο συνδέεται απευθείας με την Ασία και το Αφγανιστάν, αλλά και την Νότια, Νότιο Ασία και Φιλιππίνες και εκεί υπάρχουν προβλήματα που συνδέονται άμεσα με τον ISIS. Επομένω, ε, αυτό το πρόβλημα δεν θα λυθεί σύντομα. Για το Αφγανιστάν έχετε δίκιο. Υπάρχει σημαντικός προβληματισμός στη διεθνή κοινότητα για την κατάσταση εκεί, αλλά και για την πολιτική κατάσταση. Ξέρετε ότι ε, είναι αλληλένδετα αυτά τα δύο. Η επιτυχία στο Αφγανιστάν, μεταξύ άλλων, βασίζεται και σε ένα εύρυθμα λειτουργών πολιτικό σύστημα. Και αυτό δεν είναι εύκολο για όσους κατανοούν την κατάσταση στο Αφγανιστάν. Δεν είναι εύκολο λοιπόν να επιτευχθεί. Υπάρχουν ορισμένες εντάσεις. Υπάρχει βέβαια και πρόοδο σε στρατιωτικό επίπεδο σε ορισμένες περιοχές, αλλά και δυσκολίες σε ό,τι αφορά την πρόοδο των Ταλιμπάν τη στρατιωτική. Προβληματισμό υπάρχει και για τον ISIS και την παρέμβασή του εκεί και εδώ υπάρχουν πολλέ επιμέρου απαντήσει. δεν μπορώ εγώ να σα πω δηλαδή συγκεκριμένα. Με μεγάλη προσοχή θα πρέπει να εξετάζουμε το Ουσμπεκιστάν γιατί υπάρχει εκεί ένα φαινόμενο αλλοδαπών μαχητών από το Ουσβεκιστάν, περίπου 500 μάλιστα. ένα από αυτού ήταν ανάμεσα ε, στου τρομοκράτε στο Παρίσι. Δεν γίνεται πιο σταθερή απαραίτητα η κατάσταση. Αλλά έχετε δίκιο. Η συμμαχία ποτέ δεν έχει θέσει χρονοδιάγραμμα για, τον, για το Resolute Support Mission, γιατί δεν μπορεί να τεθεί τέτοιο όριο, θεωρούμε. Βρισκόμαστε σε μία καθοδική ε, πορεία σε ό,τι αφορά ε, τις μεταφερόμενες στρατιωτικές δυνάμεις. Θέλαμε να το σταματήσουμε, λοιπόν, ε, κυρίως ο πρόεδρος Ομπάμα, γιατί είχαν αλλάξει συνθήκες και δεν θεωρούσαμε ότι οι αφγανικέ ε, δυνάμει ασφαλείας αν μπορούσαν να χειριστούν πλήρω την κατάσταση. Εξετάζουμε τώρα τι συμβαίνει, αξιολογούμε την κατάσταση και είναι δεδομένο ότι η επόμενη προεδρική αρχή στις ΗΠΑ θα εξετάσει με μεγάλη προσοχή την κατάσταση στο Αφγανιστάν. Επομένω, ε, τηρούμε στάση αναμονή εδώ, γιατί μέχρι το επόμενο καλοκαίρι θεωρώ, παρότι δεν έχω πληροφορίε εκ των έσω, θεωρώ ότι θα υπάρξει μια αναθεώρηση από τον επόμενο πρόεδρο ε, σε ό,τι αφορά την κατάσταση στην, ε, το Αφγανιστάν. Και βεβαίω τον ΝΑΤΟ με μεγάλο μεγάλο ενδιαφέρον θα περιμένει τα αποτελέσματα. Αποφασίσαμε όμω, κλείνοντα για το Αφγανιστάν, στη Βαρσοβία, να συνεχίσουμε τη χρηματοδότηση με πολλά δις ευρώ ε, προσπάθειες ε, στο Αφγανιστάν. Για το Ιράκ μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα αυτά τα θέματα της ε, κατάρτισης, ε, της εκπαίδευσης, γιατί ακριβώς προσπαθούμε να βελτιώσουμε την εκπαίδευσή μας. Εγώ πήγα στο Ιράκ ε, ορισμένες φορές πρόσφατα και εγώ έθεσα το ερώτημα γιατί δεν πήγαν καλύτερα τα πράγματα στο παρελθόν και τι πρέπει να αλλάξουμε για να πάνε τα πράγματα καλύτερα αυτή τη φορά. Εν μέρη η απάντηση ήταν η θεσμική αναθεώρηση μεταρρύθμιση μάλλον. Να έχουμε λοιπόν ένα σύστημα θεσμικά όργανα που να λειτουργούν καλά από μόνα τους. Να μην χρειάζεται η εξωγενής παρέμβαση. Συνδέουμε λοιπόν τις προσπάθειες που καταβάλουμε εμείς προς την θεσμική μεταρρύθμιση ε, για να συνεχίσουν μετά τα πράγματα από μόνα τους. Βέβαια, ξέρετε, ε, στο Ιράκ ότι υπήρξαν και ζητήματα πολιτικά, με τον κύριο Αλμάλικη, δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε όλα αυτά βεβαίως. Εμείς ελέγχουμε ε, τη συνδρομή που παρέχουμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και την άμυνα. Να πω τα εξή. Είναι και οι λόγοι για του οποίου οι σύμμαχοι πήραν τι αποφάσει που πήραν σε ό,τι αφορά το συντονισμό με την Ένωση αν δείτε αρχικά τις υβριδικές απειλές. Για την υπεράσπιση των κρατών μελών μας, ε, το ΝΑΤΟ είναι ιδιαίτερα ισχυρό σε ορισμένες περιοχές και όχι τόσο ισχυρό ε, σε άλλες και αυτά λειτουργούν συμπληρωματικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν εξετάσουμε λοιπόν μια ευρυδική απειλή σε μια ε, χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ μπορεί να συμπεριλαμβάνει όλα τα στοιχεία αυτά ε, της ε, επίθεσης στον κυβερνοχώρο, στρατηγικές ε, επικοινωνίες αλλά και πραγματικές, στρατοτικέ, δηλαδή πλέον, απειλές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από μόνη της δεν μπορεί να παράσχει επαρκή κάλυψη και στήριξη προς ε, ένα κράτος μέλος, ούτε το ΝΑΤΟ. Από κοινού όμως μπορούμε. Ε, στις υβριδικέ απειλές λοιπόν έχει νόημα να συνεργαστούμε. και είπε και ο συνάδελφο ότι υπάρχουν συγκεκριμένε προσπάθειε και θέλουμε να λειτουργούν συμπληρωματικά. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την οικοδόμηση δυναμικού, πόσου δηλαδή, πόσε δυνάμει έχουμε εμεί στην Ουκρανία και πόσου έχετε εσεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δείτε και τα ποσά που δαπανώνται, λογικό είναι να μην ε, ε, επαναλαμβάνουμε τα ίδια και τα ίδια, ούτε να δαπανούμε ποσά μάταια. Και πολλές φορές ε, υπάρχει σύγχυση και επιτόπου, δηλαδή από αυτούς που δέχονται τη βοήθειά μας, ε, ως προς τι να, κάνουν. Τώρα για την Τουρκία, είναι βεβαίω λεπτό το ζήτημα, το είπατε κι εσείς. Να πω όμως το εξής, Όλοι οι σύμμαχοι αναγνωρίζουν πρώτα απ' όλα πόση πίεση δέχεται η Τουρκία από τη γειτονιά της. Γιατί φιλοξενεί 3 εκατομμύρια πρόσφυγες σε μία μόνο χώρα, έτσι. Και δεν πρόκειται μόνο για πρόσφυγες που έρχονται από ε, μακριά. Πρόκειται για έναν πόλεμο ακριβώ δίπλα τους, στην πόρτα τους. Αντιμετωπίζουν προβλήματα τρομοκρατίας και μια σύνθετη εσωτερική κατάσταση που συμπεριλαμβάνει και ένα, ένα πραξικόπημα ή μια απόπειρα πραξικοπήματος ε, πρόσφατα με όλες ε, τις επιπτώσεις αυτού. Αναγνωρίζουμε λοιπόν όλη αυτή την κατάσταση. Έχετε ακούσει και τον προβληματισμό σε ό,τι αφορά την αντίδραση σε αυτό το πραξικόπημα, ότι θα πρέπει δηλαδή και αυτό να γίνεται σύνομα ακόμα και στην Ιατουρκία. Έχουμε λάβει γραπτές διαβεβαιώσεις από πλευράς ε, της Τουρκίας ότι ε, θα λειτουργήσουν, ε, θα ενεργήσουν σύνομα. Είμαστε σε επαφή και από τότε με τους επικεφαλείς με τους ηγέτες δηλαδή αυτής της χώρας και έτσι στηρίζουμε ε, τα θεσμικά όργανα, του δημοκρατικού θεσμούς ε, της Τουρκίας. Χαιρόμαστε ιδιαίτερως που δεν ανατράπησαν και χαιρόμαστε που οι ηγέτες έχουν ε, αναλάβει τη δέσμευση να ενεργήσουν ε, νόμιμα. Συγγνώμη που μακρηγορώ, αλλά θα σας διευκολύνω και εσάς στην πορεία. Για τα AWACS, πραγματικά δεν γνωρίζω την απάντηση. Μπορώ να σας πω πολύ σύντομα λοιπόν ότι δεν γνωρίζω πότε θα υλοποιηθεί. Ρωσία. Μέτρα για τη διαμόρφωση ενός κλίματος εμπιστοσύνης. Νομίζω ότι το σημείο εκκίνησης για του συμμάχους είναι ότι αφενός εμείς δεν διαμορφώσαμε τις προποθέσει υπονόμευση της εμπιστοσύνης. Επομένω, είναι λάθος να δημιουργήσουμε την εντύπωση ότι τώρα είναι δική μας κυρίαρχη ευθύνη να αποκαταστήσουμε τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ευρώπη και αν αυτό δεν συμβεί αυτό είναι επειδή εμεί δεν ενεργήσαμε αρκετά εφάνταστα ή ανοιχτά. Είναι πραγματικότητα, είναι γεγονός ότι η Τουρκία εισέβαλε σε γειτονική της χώρα, ε, έχει προσαρτήσει εδάφη αυτής της χώρας και το καθεξής. Όμως εμείς θέλουμε να είμαστε ανώτεροι, να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, να αρχίσουμε ένα διάλογο και αν αυτός είναι επικοδομητικός, ενδεχομένως σιγά σιγά να πάρουμε και άλλα μέτρα για να ενισχύσουμε την προβλεψιμότητα και τη διαφάνεια στην Ευρώπη. Ακριβώς από εκεί θέλουμε να ξεκινήσουμε. Διαφάνεια και προβλεψιμότητα. Τουλάχιστον να έχουμε αυτά τα δύο. Όμως και αυτό δεν είναι απλή υπόθεση. Σας το λέω ανοιχτά. Γιατί κάποιος νομίζω αναφέρθηκε στις ασκήσεις SNAP. Δεν θυμάμαι ποιος. Οι ασκήσεις SNAP που έχει υιοθετήσει πλέον η Ρωσία ως μέσο ασκήσεων είναι εξαιρετικά αποσταθεροποιητικές γιατί κινητοποιούν συστηματικά ε, χιλιάδες στρατιωτών και στα σύνορα με τους συμμάχους μας χωρίς καμία προειδοποίηση και χωρίς σχεδόν καμία εξαίρεση ε, αναφέρουν μικρό τους αριθμούς ε, στρατιωτών στις μετακινήσεις και έτσι ξεφεύγουν από τις νόμιμες υποχρεώσεις τους υπό τη Συμφωνία της Βιέννης για να επιτρέψουν επιθεωρήσεις. Αυτό συμβαίνει ξανά και ξανά, για να αποφύγουν δηλαδή τους ελέγχους. Και αυτό δημιουργεί σημαντική αβεβαιότητα στις γειτονικέ χώρες. Υπάρχουν λοιπόν πολύ απλά και εύκολα βήματα που θα μπορούσε να αναλάβει η Ρωσία για να αποκαταστήσει αυτό το κλίμα εμπιστοσύνη, να ακολουθήσει τις υποχρεώσεις ε, που έχει αναλάβει και πιο συγκεκριμένα από το έγγραφο της Βιέννης. Παρ' όλα αυτά η Ρωσία δημοσίως έχει ε, κάνει προτάσεις για πιθανές συζητήσεις, για την ασφάλεια ε, στον αέρα, ιδίω στη Βαλτική. Περαιτέρω συζητήσεις κειμένους τομείς. Θα εξετάσουμε όλα αυτά με μεγάλη προσοχή λοιπόν και θα απαντήσουμε στην Ρωσία όμως με τα όσα εμείς ως σύμμαχοι θα θέλαμε να δούμε, να ελοποιούνται για να ε, αυξηθεί και να βελτιωθεί η προβλεψιμότητα και διαφάνεια. Και μάλιστα αυτή η απάντηση θα έρθει με σε επόμενε εβδομάδε. Υπάρχει λοιπόν ε, εσωτερικά στο ΝΑΤΟ ένα τέτοιο διάλογο. Κάποια στιγμή ελπίσουμε και με τη Ρωσία. Και να πω και κάτι με τη, για τη Φιλανδία και τη Σουηδία, γιατί έχουν ε, βρεθεί ε, στη μέση, είτε το θέλουν είτε όχι. Ε, πρέπει να αποτελέσουν τμήμα της λύσης γιατί είναι πολύ σημαντικοί σύμμαχοι. Γι' αυτό πρέπει και αυτοί να συμβάλλουν. Τέλος, ό,τι αφορά την Ουκρανία. Το Βαρτολωτικό Συμβούλιο θα μεταβεί ε, στη Γεωργία μεθαύριο με επικεφαλή στο Γενικό Γραμματέα. Είναι η τέταρτη επίσκεψη του Συμβουλίου στη Γεωργία και θα εξετάσουν ε, με μεγάλη προσοχή ε, την υλοποίηση του πακέτου, όπως αποκαλείται, για να υπάρχει μεγαλύτερη παρουσία του ΝΑΤΟ στη Γεωργία, αλλά και της Γεωργίας στο ΝΑΤΟ αύξηση και ενίσχυση των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων, των ασκήσεων. Η Γεωργία είναι και από τους μεγαλύτερους συμβολείς στις ε, στρατιωτικές επιχειρήσεις μας στο Αφγανιστάν. Αποτελεί τμήμα των ε, δυνάμεων ανταπόκρισης ε, του ΝΑΤΟ. Συνεργάζονται πολύ στενά μαζί μας και βεβαίως φιλοδοξούν να προσχωρήσουν και στο ΝΑΤΟ. Και για την Ουκρανία βέβαια είναι η εκτίμηση, μια πρόσφατη εκτίμηση ότι το 80% των παραβιάσεων ε, της ε, εκεχηρίας ε, προκύπτουν από τους μαχητές, αγωνιστές, αποσχιστές ανάλογα με το φορέα. Υπάρχει όμως μια επιδείνωση ό,τι αφορά το, το κλίμα. Το ΝΑΤΟ θέλει να στηρίξει την Ουκρανία σε ό,τι αφορά την οικοδόμηση θεσμών μακροπρόθεσμα. Όμως θέλουμε να αντιμετωπίσουμε και τις πιο βαρχιπρόθεσμες επιπτώσεις, στρατηγικές επικοινωνίες για παράδειγμα, για να αντιμετωπίζουν ε, τις υβριδικές ε, απειλές στην επικοινωνία, αλλά και στήριξη προς ε, τα θύματα, Προσπάθησε ότι αφορά την εξουδετέρωση ναρκών, και το καθεξής. Θέλουμε όμως μακροπρόθεσμα ε, να διαμορφώσουμε ένα θεσμικό πλαίσιο. Μακρηγόρησα, όντως, λέει ο συνάδελφος. Ο κύριος Φώστερ. Ναι, ο Τζέιμς μακρηγόρησε. Δεν έχουν μείνει και πολλά σημεία για μένα, αλλά με τα χαράς να σας τα σχολιάσω. Καταρχάς, κύριε Γκάλερ, η πρόταση να δεσμευτούν κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για να, την ανοικοδόμηση της Ανατολικής Ευρώπης θα το σχολιάσει ο συνάδελφος κατά πόσον προβλέπεται αυτό ή όχι, γιατί θεωρώ ότι είναι εξαιρετική ιδέα. Ε, καταρχάς γιατί έχουμε πολλά να κάνουμε και δεύτερον ε, το μεγαλύτερο τμήμα αυτών το οποίο πρέπει να γίνουν στην Ανατολική Ευρώπη δεν είναι στρατιωτικές υποδομές, είναι πολιτικές υποδομές αναφερθήκατε σε κάτι πολύ απλό, αεροπορικούς διαδρόμους. Αν θέλουμε να πετάξει η VJTF, η ομάδα απάντησης του ΝΑΤΟ, πρέπει να πετούν με F-17. Ε, Οι περισσότεροι διάδρομοι στην... σε 17, συγγνώμη. Οι περισσότεροι διάδρομοι λοιπόν δεν αντέχουν τέτοιες υποδομές. Πρέπει λοιπόν να γίνουν αρκετές επενδύσεις και εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να διαθέσει κονδύλια γι' αυτό, θεωρώ ότι είναι εξαιρετική ιδέα. Και ε, σε μεγάλο βαθμό απαντά και στην ερώτηση του κυρίου Βανόρδεν. Πού θα ήταν χρήσιμο να συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να συμπληρώσει αυτά τα οποία κάνει το ΝΑΤΟ. Αυτό είναι εξαιρετικό παράδειγμα. Ε, παρεμπιπτόντως δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όσο σκέφτεστε εσείς. Σε όλη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή οι υποδομές δεν είναι στα χέρια των κρατών οι υποδομές σε μεγάλο βαθμό είναι ιδιωτικοποιημένες και στα χέρια ιδιωτικών επιχειρήσεων και σε πολλές περιπτώσεις ούτε καν επιχειρήσεις ε, ε της χώρας. Μπορεί να είναι οι επιχειρήσεις από τρίτες χώρες, μπορεί και ρώσικες. Να σας δώσω το παράδειγμα. Το μεγαλύτερο λιμάνι της ε, Μεσογείου, ε, ο Πειραιάς στην Αθήνα, είναι κινέζικης ιδιοκτησίας. Όλα αυτά περιπλέκουν τα πράγματα, αλλά η ιδέα αυτή καθεαυτή ε, θα μπορούσα κάλλιστα να την υποστηρίξω. Και φυσικά η άμυνα είναι πολύ δαπανερή η υπόθεση και το θέμα της στέγασης των στρατευμάτων μπορεί να είναι απλώς ψήγμα των όλων δαπανών. Ο Τζέιμς αναφέρθηκε στην άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από πλευράς παραδοσιακής πολιτικής άμυνας, που είναι η δική μου αρμοδιότητα. Αυτό το οποίο διαπιστώνω είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπε και ο Τζέιμς, έχει διαφορετικά εργαλεία τα οποία ε, χωρούν στην ίδια εργαλοθήκη και χαίρομαι που μπορούμε να τα ε, χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά από κοινού και από ό,τι βλέπω, σε πολλέ περιπτώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαφορετικέ προτεραιότητε από το ΝΑΤΟ. Εντάξει, η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν μπορεί να κάνει αυτό που θέλει, επικεντρώνεται σε άλλου τομεί, σε άλλα μέρη του κόσμου. Και πάλι τώρα όσον αφορά ε, τη συμπληρωματικότητα, αν κάνω λάθος διορθώστε μου, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ε, περίπου 70 αποστολές και επιχειρήσεις και πραγματικά δεν νομίζω ότι υπάρχει ανταγωνισμό στον τομέα. Ε, λειτουργεί πολύ αποτελεσματικά το σύστημα και Εκεί που υπάρχει θέμα είναι φυσικός καταμερισμός εργασίας. Ε, ο ένας οργανισμός επικεντρώνεται στο ένα σημείο και ο άλλος στο άλλο. Ε, δεν είναι άσπρο-μαύρο τα πράγματα, αλλά όσον αφορά την έκδοση κοινών δηλώσεων είναι ένας φυσικός τρόπος λειτουργίας των πραγμάτων. Όσον αφορά την Τουρκία δεν νομίζω ότι να νομίζουμε ότι ο Νότος διαφέρει εξ ολοκλήρου με το Βορρά ή με την Ανατολή. Οι δύο περιοχές της Ευρώπης έχουν διαφορετικά προβλήματα και δεν είναι αλληλένδετα. Απλώς πρέπει να συνειδητοποιήσετε τώρα ότι η Τουρκία έχει ρωσική στρατιωτική παρουσία σε τρεις πλευρές. Έχουν τους Ρώσους στην Κρυμαία, η Γεωργία και στη Συρία. Επομένως αυτά συνδέουν το πρόβλημά τους, αλλά από την άλλη ως σύμμαχος του ΝΑΤΟ ε, είναι πάρα πολύ σημαντική και για τα όσα ε, συμβαίνουν βορειοανατολικά. Υπήρξαν κάποιες ερωτήσεις από τον κύριο Ζήμ και δεν ξέρω αν προφέρω σωστά το όνομά σας. Καταρχάς, όσον αφορά την Πολωνία και το ρόλο της ως ε, ε, Συνόδου. Ήταν εξαιρετική η σύνοδος κορυφή όσον αφορά την διοργάνωση, την ασφάλεια. Τα πράγματα ήταν εξαιρετικά και νομίζω ότι τα συγχαρητήρια ακούστηκαν από όλου ε, προς την πολωνική κυβέρνηση για την ε, πάρα πολύ καλή διοργάνωση. Τα πάντα ήταν εξαιρετικά. Το κατά πόσον η στρατιωτική απάντηση δεν επαρκεί, αυτές οι μονάδες μάχης που αναφέρατε, είναι σαφώς ε, μεγαλύτερες τάγματα, αλλά να σας το πω εξής η ενισχυμένη ε, παρουσία, αυτές οι μονάδες μέχης που ε, συστήνουμε είναι απλώς ένα τμήμα της στρατιωτικής μας ε, παρουσίας. Τα ε, έχουμε σε τρία σκέλη αυτό. Το πρώτο σκέλος αφορά τις δικές σας δυνάμεις άμυνας και για την Πολωνία σε καμία περίπτωση δεν είναι ελάχιστες. Είναι τεράστιες, έχουν εξαιρετικές δυνατότητες και μπορούν σε πολύ μεγάλο βαθμό να υπερασπιστούν και τη χώρα αλλά και τις γειτονικές σας χώρες. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος. Οι ε, μονάδες μάχης ε, οι οποίες συστήλουμε αυτά τα τέχματα ε, θα έρθουν να ενταχθούν στις εθνικές σας ενόπλες δυνάμεις. Για τα χώρες της Βαλτικής ο στρατός είναι λίγο μικρότερος αλλά δημιουργούν σε μεγάλο βαθμό και τις δικές τους τις ενόπλες δυνάμεις. Αυτά λοιπόν είναι η πρώτη κλίμακα. Η δεύτερη κλίμακα είναι η ομάδα απάντησης του ΝΑΤΟ. Ε, η δύναμη αυτή αυτή τη στιγμή αριθμεί 40.000 στρατιώτες και μπορεί να απαντήσει εντός ημερών και σας διαβεβαιώ είναι καθόλου ικανή και μπορεί και να αυξηθεί το πρώτο σκέλος ε, μπορεί να κινητοποιηθεί πολύ γρήγορα αν χρειαστεί είτε για αποκλιμάκωση μιας κρίσης είτε για μάχη εάν χρειαστεί. Και το τρίτο σκέλος είναι η δυνάμεις που ακολουθούν όπως τι αποκαλούμε. Είναι περίπου 2.000 ε, άνδρες ή γυναίκες σε χώρες του ΝΑΤΟ. Εάν λοιπόν τα προσθέσετε αυτά τα τρία και τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται, ε, τοποθετούνται και κάνουν και τις ασκήσεις τους, οι μονάδες μάχης είναι σημαντικές, είναι ε, δύναμη κρούσης, αλλά είναι ένα μικρό τμήμα της ευρύτερης εικόνας. Αναφερθήκατε σε πολλαπλές εθνικότητες για το κατά πόσο χρειαζόμαστε διερμηνείς και μεταφραστές. Ε, δεν ε, θα σας κρύψω ότι το γεγονός ότι είναι πολυεθνικές αυτές οι ομάδες, ιδέως ε, σε κατώτερο επίπεδο, ε, μπορεί να ε, έχετε λίγο να ε, υποδυναμώσει τις δυνατότητες μάχης, αλλά αυτό το πολυεθνικό στοιχείο είναι πολιτικό αγαθό, γιατί αν θέλουμε να έχουμε το άρθρο 5 και να υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ των συμμάχων, πρέπει να υπάρχει παρουσία ε, πολυεθνική ε, ομάδες από διάφορες εθνικότητες, συμπεριλαμβανομένων και των Ηνωμένων Πολιτειών φυσικά. Και παρά το γεγονός ότι είναι επικεφαλή σε μία από τις τέσσερι μονάδε μάχη, έχουν παρουσία σε κάθε χώρα, σας διαβεβαιώ. Για τις ασκήσεις SNAP ε, υπάρχουν ε, μεγάλες κινητοποίησεις ε, στην ανατολική πλευρά των συνόρων μας. Ο James αναφέρθηκε στο θέμα αυτό ήδη. Εμείς ε, δεν κάνουμε κάτι αντίστοιχο για αρκετούς λόγους. Πρώτον και κυριότερον γιατί έχουμε αμυντικούς σκοπούς και όχι επιθετικούς σκοπούς. Αν γίνεται τέτοια κινητοποίηση τότε σαφέστατα έχεις επιθετικές προθέσεις. Ε, δεν γίνεται λοιπόν κάτι τέτοιο. Δεύτερον, δεν θεωρούμε ότι έχουμε ψυχρό πόλεμο αυτή τη στιγμή, όπως ε, πριν από 25 χρόνια. Και δεν πρόκειται να ε, στήσουμε απέναντι στα στρατεύματα αυτά, τα δικά μας στρατεύματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε δυνατότητα απάντηση σε αυτές τις κινήσεις. Υπάρχουν διάφορες δυνατότητες απάντησης, τις οποίες δεν θα σας αναφέρω εδώ, αλλά ε, σε καμία περίπτωση ε, δεν θα βρεθούμε προεκπλήξεων. Και αυτό με φτάνει και στην τελευταία ερώτηση του κ. Φρόιντ πόλεμο στην Ευρώπη. Ο ψυχρός πόλεμος ε, ήθελε σε μεγάλο βαθμό να προλάβει ε, πόλεμο στην Ευρώπη, αλλά αν χρειαστεί θα μπορούσε να γίνει και η μάχη. Με μια Ρωσία τώρα που θεωρούσαμε, ε, θεωρούμε στρατηγικό εταίρο, έχουμε σαφώς ξεφύγει από την ιδέα ότι θα πρέπει ε, να υπερασπιστούμε την Ευρώπη. Τώρα πλέον με μια επιθετική Ευρώπη η οποία έχει βάλει σε σύνορα σε γειτονικέ μας χώρες και έχει απειλήσει ε, κάποιους από τους συμμάχους ε, του ΝΑΤΟ είτε λεκτικά είτε και μέσω κινήσεων στα σύνορα και με δηλώσεις του Πούτιν για αυτές τις κινήσεις δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε αυτές τις εξελίξεις και πρέπει να είμαστε σε θέση να υπερασπιστούμε την Ευρώπη εάν τα πράγματα φτάσουν τα άκρα. Γι' αυτό ακριβώς και στην ε, Σύνοδο της Βαρσοβίας ε, έχουμε μία σειρά από μέτρα ε, τα οποία πρωτίστως στόχο έχουν την πρόληψη οποιασδήποτε αντιπαράθεσης, είτε στρατιωτική είτε πολιτικά μέτρα, αλλά εάν φτάσουν τα πράγματα στα άκρα και πρέπει να γίνει πόλεμος, ε, τότε θα πολεμήσουμε. Ελπίζουμε περιορισμένους και για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά ε, κάνουμε προσαρμογές από στρατιωτική σκοπιά ε, για να μπορέσουμε να κινηθούμε σε όλη την Ευρώπη. Και αυτό συνδέεται με όλα αυτά τα πράγματα. Και νομίζω ότι με αυτό κάλυψα όλα τα σημεία. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ και εσάς. Κύριε Κλόντι, σειρά σας να απαντήσετε στις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Βρίσκομαι σε πολύ εύκολη και ευχαριστή θέση, διότι ήδη απαντήθηκαν από τους συναδέλφους οι περισσότερες ερωτήσεις. Και σίγουρα δεν πρόκειται να διαφωνήσω με αυτά που είπαν. Να επανέλθω στις τελευταίες δύο ερωτήσεις που έγιναν. Η ερώτηση του κυρίου Γκάλερ για πιθανότητα στήριξη από τον Ευρωπαϊκό προπολογισμό στις υποδομέ υποδομές μας. Νομίζω ότι μου απάντησε σε αυτό, αλλά εάν πρόκειται για πολιτικές υποδομές σε μια χώρα εταίρο, τότε σίγουρα η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη έχει στηρίξει αυτές τις προσπάθειες και μάλιστα με δισεκατομμύρια ευρώ. Το πρόβλημα αρχίζει όταν η υποδομή είναι στρατιωτική ή έχει αμυντικό χαρακτήρα. Εδώ μπορώ να σας ε, δώσω πολλά παραδείγματα, τα οποία δείχνουν ότι παρά τις ε, μεγάλες ανάγκες που υπάρχουν για να γίνει κάτι τέτοιο, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Και ε, ένας από τους τρεις στόχους, μία από τις τρεις προτεραιότητες μάλιστα της πολιτικής μας είναι και η δημιουργία ικανοτήτων. Δεν μπορούμε ακόμα να το κάνουμε πράξη αυτό, διότι ο αποδέκτης είναι ένας διαφορετικός στρατιωτικός οργανισμός. Κάτι που ήδη αναφέρθηκε στην Επιτροπή εδώ. Γι' αυτό λοιπόν κολλιόμεθα. Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός δεν μπορεί να στηρίξει κάτι τέτοιο. Εκτός μικροφώνου το σχόλιο του κυρίου Γκάλερ. Ακριβώς, λέει ο κύριος αυτό είναι το ζητούμενο. Η ερμηνεία δηλαδή πώς να ερμηνεύσουμε το άρθρο 41.2 της ε, συνθήκης. Αυτός λοιπόν ήταν και ο σκοπός για τον οποίο ε, συντάχθηκε αυτό το άρθρο, δηλαδή να στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις. Όταν όμως ε, το ζητούμενο είναι η δημιουργία ικανοτήτων, η Ευρωπαϊκή Ένωση το κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες. Βοηθά τις χώρες να δημιουργήσουν τις κατάλληλες υποδομές, τις κατάλληλες ικανότητες. Εκεί μπορούμε να βοηθήσουμε. 80 δισεκατομμύρια ευρώ δαπανήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση το περασμένο έτος σε τέτοιες ε, υποδομές. Δεν γίνεται όμως να χρησιμοποιήσουμε κονδύλια από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό, τα οποία θα πάνε σε έναν ξένο στρατιωτικό οργανισμό. Αυτά ως προς αυτό το θέμα. Είναι όντως ένα πρόβλημα. Ένα άλλο πρόβλημα σχετικό με αυτό είναι ότι πολλές φορές ε, δυσκολευόμαστε να χρηματοδοτήσουμε τις δικές μας δραστηριότητες. Αυτό δηλαδή που έχετε ακούσει ως 10% αλληλεγγύη, 10% μόνο του ε, κόστους ε, για κάτι είναι κοινό ή θεωρείται κοινό. Τα πράγματα όμως στο ΝΑΤΟ είναι πολύ διαφορετικά. ιδιαίτερα όσον αφορά τις ε, ομάδες μάχης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ τα θέματα ε, είναι άλλα και πρέπει να επιληθούν τα προβλήματα το προχωρήσουμε. Τώρα, το θέμα δεν είναι μόνο πόσα χρήματα μπορούμε να βάλουμε στην άκρη για να στηρίξουμε αυτά τα προγράμματα, αλλά τι μπορούμε να ξοδέψουμε και πώς μπορούμε να ξοδέψουμε τα χρήματα που διαθέτουμε. Να αναφέρω πολύ σύντομα ότι χρειάζεται να χρησιμοποιούμε τις ικανότητες που ε, διαθέτουμε και αυτές να συντηρούμε. Και εδώ έχετε κι εσείς να παίξετε, οι ευρωβουλευτές, έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Η Ευρώπη έχει ανάγκη να διατηρήσει τις υφιστάμενες ικανότητες, ποιες είναι οι προτεραιότητες, οι αμυντικές υποδομές ή οι θέσεις απασχόλησης. Αυτή λοιπόν είναι η μεγάλη πρόκληση, είναι το να ερώτημα και ε, αυτό θα προσπαθήσει να κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση με το e UGS. Και ο Τίμο αναφέρθηκε και στο αποτέλεσμα, ότι δεν αρκούν δηλαδή μόνο οι ικανότητες, δεν πρέπει μόνο να έχουμε τις δυνατότητες για κάτι, πρέπει να τις χρησιμοποιούμε και όλες. Τώρα, αντιμετωπίζουμε και εμείς τις ίδιες δυσκολίες παντού στην επικράτειά μας. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω πως τα προβλήματα είναι λίγο πολύ κοινά. Όσον αφορά τώρα το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην άμυνα, νομίζω πως με κάλυψαν οι συνάδελφοι. Αυτό που θα ήθελα ίσως να προσθέσω είναι ότι όταν κάνουμε λόγο για άμυνα, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι έχει φτάσει η στιγμή να εξυγχρονιστεί ε, η άμυνα, να επικαιροποιηθεί ο ορισμός της, γιατί η άμυνα δεν έχει να κάνει μόνο με ε, στρατιωτικό χαρακτήρα. Βέβαια, αναφέρθηκε και η διαδικασία DPPR, αλλά έχει να κάνει και με τη συλλογή πληροφοριών, έχει να κάνει με το πώς χρησιμοποιείς τις υποδομές σου, τις ικανότητες που έχεις. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω δίχως αμφιβολία, έχει συνεισφέρει σημαντικά σε αυτό. Επίσης, αναφέρατε την ανθεκτικότητα Εάν θέλουμε οι υποδομές μας και η κοινωνία μας να είναι ανθεκτική στις εξωτερικές επιθέσεις, τότε στο χέρι της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να γίνει αυτό. Για παράδειγμα, δείτε τι δύναμη έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις οδηγίες της, κάτι που δεν έχουν οι άλλοι ε, διεθνείς οργανισμοί. Βέβαια και το ΝΑΤΟ έχει κάποιες ε, δυνατότητες, όμως δεν είναι ε, το ίδιο αποτρεπτικές με τις δυνατότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρώσεις, για παράδειγμα. Οι κυρώσεις έχουν αποτέλεσμα. Όλα αυτά λοιπόν τα μέσα είναι στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω όλων αυτών να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στον τομέα της άμυνας. Σίγουρα θα ήταν ιδανικό να υπήρχε ένας οργανισμός και όχι δύο και να μην ε, υπήρχαν αυτές οι διαφορές. Σίγουρα αντί για 28 ε, αρχηγούς επιτελείου, 28 υπουργούς άμυνας, να, θα ήταν καλύτερο να υπήρχε ένας μόνο, αν ακολουθήσουμε την ίδια λογική. Όμως αμφιβάλλω για το αν αυτό είναι κάτι που θέλει έστω και ένας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή όμως είναι η πραγματικότητα που έχουμε στα χέρια μας. Έχουμε διαφορετικές χώρες, έχουμε δύο διαφορετικούς οργανισμούς και αυτό που χρειάζεται είναι να δούμε πού συμπληρώνει ο ένας οργανισμός των άλλων, πού μπορούμε να συνεργαστούμε, πώς μπορούμε να να συνεργαστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πώς δηλαδή θα χρησιμοποιήσουμε με το βέλτιστο τρόπο τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Αναμένεται να υπάρχει αγαστή συνεργασία. Αυτά προς το παρόν από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι έχει τελειώσει ο χρόνος μας, λυπάμαι πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους διακεκριμένους μας ομιλητές για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή παρουσίαση, αλλά και τις απαντήσεις τους που ήταν πληρέστατες. Σας ευχαριστώ πολύ. Αποχαιρετούμε λοιπόν ε, τους καλεσμένους μας, αλλά μπορείτε να μείνετε ε, δύο λεπτά ακόμα. Okay. Ladies and gentlemen. Κυρίε και κύριοι, θα πρέπει να εγκρίνουμε τα πρακτικά των προηγούμενων συνεδριάσεων. Δύο συνεδριάσεις της Υποεπιτροπής ε, Ασφάλειας και Άμυνας. Το παραλείψαμε στην αρχή της συνεδρίασης. Έχουμε λοιπόν τα πρακτικά της 30 Ιουνίου. και της 13ης Ιουλίου. Έλλειψη σχολείων, νομίζω ότι... Α, νομίζω πρέπει να αφήσουμε ένα περιθώριο μέχρι την επόμενη συνεδρίαση για υποβολή τυχών ε, σχολείων και επιφυλάξεων. Εάν δεν υπάρχει κάτι μέχρι τότε, λοιπόν, θα θεωρήσουμε ότι έχουν εγκριθεί τα πρακτικά. Η επόμενη συνεδρίαση και πάλι μισή μέρα θα διαρκέσει στις 26 Σεπτεμβρίου. Ωραία, τα λύσαμε και αυτά. Υπό τα διάφορα νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο. Έχουμε πει τόσο έτσι και αλλιώς σήμερα. Σας ευχαριστώ όλους λοιπόν για την ενεργό συμμετοχή σας. Yeah. That as usual, I like to... Και όπως πάντα, ευχαριστώ και τους διερμηνείς. Καλό απόγευμα.